Could Μήπως μπορούν οι κοινωνιστές συνάδελφοι... Α, Νάτι, Νάτι, εσένα περιμέναμε Κωνσταντζα και ετοιμάζουμε σαμπάνια και για φέτος. Uh, Μήπως μπορούμε να αρχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμη μερικές ψηφοφορίες. Βρισκόμαστε στην προσθήκη 1. Για όσους έχουν κατάλογο σαν τον δικό μου, είμαστε στη σελίδα 304, τροπολογία 188, ο 1808. Συγγνώμη για τους διερμηνείς, αλλά ίσως προφέρω τους αριθμούς περίεργα, αλλά να τι να κάνω. Έτσι αυτά στις συνήθειες έχω. Λοιπόν, αρχίζουμε. Τι θέλεις Ελισάβετ, ήδη είσαι υπέρ. Ξέρω και γιατί, ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 1808 ε, υπέρ, κατά. Δυστυχώς Ελισάβετ απερίφθη. Uh, abstentions, it's, uh, false. Ήτρε um, 113 υπέρ κατά εποχές απαρρίπτεται. Το πρώτο τμήμα ήταν αυτό. Τώρα το δεύτερο τμήμα της Ήτρε 113 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Και τώρα το τρίτο τμήμα της Ήτρε 113 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Το τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Πέμπτο τμήμα της Ήτρε 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1811 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1812 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1809 καταπίπτει. Αποσύρεται. Καλά, αποσύρεται. Ε, Α, ναι, μάλιστα. 1809 υπέρ. 1809 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1810. 1815 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1813 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1814 υπέρ κατά αποχές από, εγκρίνεται. 1816 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 1817 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. Τώρα περίφ 55 πρώτο τμήμα υπέρ κατά οχές απορρίπτεται. NV54 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18, 18, 1818 υπέρ. Α, εκπίπτει το 1818. Τώρα NV54. Α, το έχουμε. NV54 υπέρ. Κατά. Οχές, απορριπτεται Απορρίπτεται. NV55 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται 1819 υπέρ κατά πουχές απαρρίπτεται κουλτ 17 πρώτο τμήμα υπέρ κατά πουχές απαρρίπτεται 1820 We vote 1820 is in favor. 1820 υπέρ, κατά, εποχές, απαρρίπτεται. Κουλτ 17, δεύτερο τμήμα. Α, έχει εκπέσει, έχει εκπέσει. 1821. Καταπίπτει. Κουλτ 17, τρίτο τμήμα. Καταπίπτει. Τραν 37, Τραν 37 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. 1822 υπέρ κατά χες απαρρίπτεται. Τραν 39, α, τραν 40 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Τραν 38 ε, υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Τραν 39 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Τραν 41 υπέρ κατά οχές απορρίπτεται. 1824 υπέρ κατά οχές απορρίπτεται. 1825 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1826 υπέρ έχει καταπέσει και 1827, 1828, 1829 απασχόλησης 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1830 κατά πίπτη, όχι, 1830 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται, κουλτ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 1831 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1833 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάλι 1833 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έμπλ 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1834 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1835 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1836 υπέρ, κατά, ποιες, εγκρίνεται. Έμπλο 223 υπέρ, κατά, ποιες εγκρίνεται. 1837 υπέρ, κατά, ποιες εγκρίνεται. Κουλτ 19 υπέρ, κατά, όχι, όχι. Α, εκπίπτει, εκπίπτει, καταπίπτει. 166 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 1838 καταπίπτει 1839 καταπίπτει έμπλο 225 καταπίπτει 1840 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1841 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1842 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1843 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 1844 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπρο 6 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. 1845 καταπίπτει, 1846 καταπίπτει και η 47. 1848 απορρίπτεται. Έμπλ 227 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 1849 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Έμπλο 228 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1850 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. Έμπλο 230 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 1852 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1851 υπέρ υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται έμπλε 231 καταπίπτει 1853 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 1854 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 1855 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 1856 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται έμπλου 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1857 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλο 234 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1858 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 235 καταπίπτει, 236, 236 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 1859 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 1861 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 1860 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, ΑΕΜΠΛ 237 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 1862 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται έμπλ 238 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 1863 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1864 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται M 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1865 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται M240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1866 καταπίπτει έμπλε 241 241 έμπλε 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1867 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1868 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1869 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1000 Α, ξανά, ξανά. 1869 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1870 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 242 υπέρ στην προσθήκη 4 είπαμε συνεχίζουμε έμπλ 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1871 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 243 όχι, α, 2.44, 2.44. Περ, κατά αποχές. Απορρίπτεται 1872 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 1873 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 1874 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 1875 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 1876 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται Ήτρε 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1877 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελείωσε και αυτό και τώρα πρέπει να σας πω το εξής. Μας δίνει εντολή αυτό για την διαπραγματευτική ομάδα. Είναι κανείς κατά. Και το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω. Τι να ψηφίσουμε για την εντολή. Μα αφού ψηφίσαμε για την εντολή διπλά θα ψηφίσουμε. Ψηφίσαμε. Μα σας ρώτησα, δέχεστε ή όχι τις τροπολογίες που δεχτήκαμε ως εντολή για τη διαπραγματευτική ομάδα με το Συμβούλιο. Σηκώστε τα χέρια όσοι το δέχεστε. Το δεχόμαστε ως εντολή λοιπόν ως εντολή. Άμα θέλετε ψηφίζουμε και χωριστά, εντάξει, γιατί όχι. Μπορεί να ψηφίσουμε άμα θέλετε. Αν νομίζετε ότι χρειάζεται και λοιπόν, Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για να δεχτούμε αυτά που δεχτήκαμε ως εντολή όμως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Μα δεν το είπα ακόμη το δεύτερο. Αυτό ήταν το πρώτο. Λοιπόν, μερικοί δεν ψήφισαν γιατί βγήκαν έξω. Αλλά θα λήξει εδώ η ψηφοφορία. 34 ψήφισαν υπέρ. Μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν, 8 ψήφισαν κατά και 2 αποχές. Και άλλο ερώτημα τώρα. ο καθορισμός της ομάδας που πρέπει και αυτόν να τον εγκρίνουμε. Προτείνω η διαπραγματευτική ομάδα και αυτό τον κανονισμό να αποτελείται από την πρόεδρο, το θεωρώ καθήκον μου, τους εισηγητάς και τον συντάκτη της γνωμοδότησης για την απασχόληση καθώς και όλους τους σκιώδης. από όλες τις πολιτικές αμάδες. Συμφωνείτε λοιπόν να είναι αυτή η διαπραγματευτική ομάδα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό. Α, ναι, ήξερα ότι θέλετε κάτι να πείτε, πέστε το μετά από αυτή την τεράστια μαραθώνια ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες και για τη συνεισφορά αλλά κυρίως για την υπομονή σας για να ε, μας δώσετε αυτή την εντολή στην Κωνσταντσα και σε μένα. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι χωρίς αυτές τις τροπολογίες και παρά αυτές τις τροπολογίες υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις από διάφορα κόμματα, περιφέρειες. Θέλουμε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Βάσει αυτών λοιπόν και της εντολής που μας δίδεται ε, ε, θα ε, διαπραγματευτούμε και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Σήμερα το πρωί ακούσαμε την Κυπριακή Προεδρία. Θέλουν οι άνθρωποι να το προωθήσουν και να ψηφίσουμε για εκείνα τα άρθρα που αφορούν τα οικονομικά και τις αιτιολογικές σκέψεις το συντομότερο. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή και στο παρελθόν άλλωστε το τελευταίο εξάμεινο κάθε μήνα ενημερώναμε βήμα προς βήμα, θα το ε, συνεχίσουμε αυτό. Ε, και ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που έκανε το προσωπικό. Χιονοστιβάδα ήταν αυτή η ιστορία των τροπολογιών. Αν δεν είχαμε τους συνεργάτες μας, τι θα κάναμε. Και για όσους διστάζετε θα σας πω ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Θα σας ενημερώνουμε με ειλικρίνεια πάντα και Τώρα αυτό που κάνουμε τι είναι. Δημιουργούμε μια κατάσταση έτσι ώστε η Επιτροπή μας εδώ ε, σε όλους τους ε, κανονισμούς και από όλες τις επιτροπές είναι η πρώτη που έχει τη διαπραγματευτική εντελή για να αρχίσει ε, τη διαπραγμάτευση. Γιατί το Συμβούλιο τι λέει, το Κοινοβούλιο είναι υπέροχο. Πάμε εκεί και συζητάμε ώρες επί ωρών. Τώρα έχουμε συγκεκριμένη εντολή για συγκεκριμένα πράγματα και Ελπίζω να συνεχίσουμε. Σήμερα το πρωί η Κωνσταντσα Κρέλα έκανε μια σύντομη εισαγωγή. Εγώ κλείνω, μιλώ και εξ ονόματο τη. Νέβη Καταφατικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξέρω ότι χαίρονται ορισμένοι, αλλά έχουμε και άλλη δουλειά ακόμα και παραμένουν παρακαλώ οι συγητές. Δεν τελειώνει εδώ αυτή η ιστορία. Μην πάτε τώρα να το διασκεδάσετε. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Την έκθεση του Γιάννου Ορμπριχτ. Μπορεί να είναι μικρότερη η έκθεση αυτή, αλλά έχει τις σελίδουλες του ο κατάλογος ψηφοφορίας. Dear can we just move to the vote on uh, committee? Uh, να περάσουμε στην επόμενη έκθεση, σας παρακαλώ πολύ, ε, που έχουμε να ψηφίσουμε. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερική Ανάπτυξης, ο συμβιβασμό 1, υπέρ, και ο Λαμπέρ και η Κωνσταντσε, σα λέω εγώ τι κάνουν οι ομάδε σα, εγκρίνεται. Ε, 119 ψηφί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στη σελίδα 7 έχουμε τον ίδιο κατάλογο όλοι, 129 ψηφί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε παρακαλώ. 131 ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία. Περσέρβει ένα από το ΕΛΚ. Δυστυχώ κάποιος αναπληρωτή να πάρει την κάρτα του από το μηχάνημα. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε πάμε στα 130 τώρα. Ψηφί πέ. Κατά. απόχε. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία, αλλά πρέπει να το ξαναελέγξουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 130. Πέρας, δεν δουλεύει και γρήγορα το μηχάνημα. Ε, απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη σελίδα 10. 1.44 υπέρ Τη 144 κατά αποχές απορρίπτεται έχω την αίσθηση 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ 148 την ψηφίσαμε. Όχι, δεν την ψηφίσαμε. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ συγγνώμη τα έχω χάσει δεν είμαστε σε 149 ναι, υπέρ κατά αποχές έλεγχος δεν καταλαβαίνω τι ψηφίζεται 149 Πέρα στις ψηφοφορίες. 25-22 εγκρίνεται. 150 υπέρ. 150 υπέρ. Ορίστε. Συγγνώμη, 52. Μα πού είναι 152. Α, όχι. Πάμε στο συμβασμό 3. Ε, ψήφι Κατά... Μη με βοηθάτε σας παρακαλώ. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 στη σελίδα 12. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 158. Ένα σοσιαλιστής ιστορία είναι πέρα αριθμός. Απορρίψετε. Ο Γιάννα Όλμπριχτ ήτανε 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. 172 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, πάμε στην 184 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψετε, 185 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψετε, 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε σας παρακαλώ πολύ. 187 δεν βλέπω από εδώ τι γίνεται. πίπτη... Όχι, καταπίπτει, αφήστε τη. Α, ήθελα να σα κοιμάσω, αν κοιμάστε, αλλά δεν αντιδράτε κιόλα. Τι να κάνω. 89. 189. Καταπίπτει 190. Όχι, μισό λεπτό. 189. Υπέρ. Mm. κατά αποχές απορρίπτεται. Μας... Now we go to 190. Who's in... 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε σας παρακαλώ πολύ την 195 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 16 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 Καταπίπτει. Και πάμε στη 202. Ψήφι υπέρ. 202. Υπέρ. Μόνο ο Λαμπέρ και ο Κέλλη ψηφίζουν. Το ΕΛΚ τι είναι, είναι υπέρ. 202. 203 καταπίπτει είπαμε. 202 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. 18. Βιομηχανία. Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209. Εκεί δεν όχι. Προτιμάει τη 227. Ό,τι μου πείτε. 227. Είναι στην άλλη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 228. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Ε, απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά Δεν εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη τροπολογία 15. Υπέρ. Συνάδελφοι, δεν σηκώνετε χέρια, δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίζετε. Κατά... Ε, και πάλι χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 7 ψήφους. Τώρα, τη 2.36 θα ψηφίσουμε. 39, συγγνώμη, 2.39 υπέρ. 2.39. Ποια ματσόνη. Τι θες Λαμπέρ, τι κάνεις. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 τη Επιτροπής Μεταφορών υπέρ. Α, όχι, είναι ταυτόσιμες, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, ζητώ συγγνώμη. 2.40 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Η συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ακολουθεί η συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Αν δεν θέλουν οι σοσιαλιστές έλεγχο, δεν τον ελέγχουμε. Τα υπόλοιπα έχουν αποσυρθεί, αποσυρθεί. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στη συμβαστική ναι, έχουμε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε πρώτα το πρώτο, ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά ελέγχουμε το πρώτο τμήμα, λέει η Πρόεδρος της Συμβαστικής Τροπολογίας του Περιφόρων ναι. Yes, yes, Κάτι δεν καταλαβαίνω. Λέει η κυρία Ντελή, αφού το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε. Ή αποσύρθηκε. Όχι, αποσύρθηκε και ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο. Ποιο είναι υπέρ του δεύτερου τμήματο, παρακαλώ λέει η πρόεδρο. στη συμβιβαστική 9. Το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε, όχι το πρώτο. Το, λοιπόν, το ψηφίσαμε το δύο, εγκρίθηκε έτσι. Και ακολουθεί. Μα δεν το ψηφίσαμε τώρα. Το δεύτερο τμήμα. Αν νόμιζα ότι το είχαμε γκρίνει. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα λοιπόν, Λάμπερτ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο πάντα τμήμα της απολογίας 9 της συμβαστικής. Μου λένε τώρα να πάω στη σελίδα 30. Αγαπάω. πάω. 271. Του κυρίου Σόνικ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τη συμβαστική υπαριθμών 11 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάλι πηδάμε αρκετέ σελίδες. Και πάμε στην 34. Η τροπολογία 292. Υπέρ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 12 σε δύο τμήματα το ψηφίζουμε και τα δύο λοιπόν πρώτο το πρώτο υπέρ στο συμβασμό 12 κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα στην τοπολογία 300 στην επόμενη σελίδα στην 36 η τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 12α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Στην 317 πάμε, σελίδα 38. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνεται χέρια. Κατά, άρα απορρίπτεται, εντάξει. Άμα απορρίπτεται, εντάξει. 318 υπέρ. 318. Είμαστε σε επόμενοι. Υπέρ, κατά. Ελέγχουμε την 318 παρακαλώ. Και απορρίπτεται. 300... Όχι, 320 μια στιγμή. Η 11 τη επιτροπή Προπολογισμού, βλέπετε λίγο πιο κάτω στη μέση τη Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψετε. Στην επόμενη σελίδα, 330 ε, υπέρ, σελίδα 39. Τι λέτε ότι έπρεπε να ψηφίσουμε την 320. Θέλετε να την ψηφίσουμε 320, καλώς. Υπέρ. Identical λέει εδώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 330. Εάν δεν κάνουμε λάθος εδώ πάνω υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε καταπέσει. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Mm. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα. 42. Σελίδα 42. 27 καταπίπτει τη Ήτρε. Η 356 τώρα, στη σελίδα 42, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 359 ψηφίστηκε. 357 υπέρ. Κατά έλεγχος για την 357. Απορρίπτεται. 358 καταπίπτει. 29 της Ήτρε όχι. 29 της Ήτρε ψηφίζουμε. Επιτροπή Βιομηχανίας. Ε, υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι στην 30 της Ήτρε είμαστε τώρα υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 361 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 368 όχι 32 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβατιστική 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 τι έγινε Α, ο συμβιβασμό εγκρίθηκε, λέει η γραμματεία. Ε, γι' αυτό πρέπει να με διορθώνετε. Ε, όταν λέω ότι απορρίφθηκε να μου το λέτε. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την 380. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 381 Κατά Ναι. 35 ήτρε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 383 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 353 Συγγνώμη, 383. Λαμπέρ, αν ήσουν και πιο θετικό στη αντίδρασή σου, θα ήταν όλα πιο εύκολα και αληθινά ίσως. Ε, κάθε φορά πρέπει να ελέγχω επειδή είστε εσείς κατά. Απορρίπτεται. 27-19. 386 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα πάμε στη σελίδα 46 και έχουμε την τροπολογία 397. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καταλήπτει. 398 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 399 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τετρακόσια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι ταυτόσημη εντάξει 401 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 405. Πρέπει να ψηφίσουμε την 405. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 403 υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. 400... Πάμε στη συμβιβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 415 υπέρ κατά ελέγχουμε 415 Απορρίπτεται. 28 τραν πηγαίνουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 39 ήτρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 4.30 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται, 44 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 416 περα κατά έλεγχος ηλεκτρονικός για την 416 Απορρίπτεται. 431. Πολλοί δεν ψηφίζουν. Κατά. Απορρίπτεται. 4,21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 4,17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4,18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4,19 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται,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 κατά αποχές απορρίπτεται 437 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 439 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 438 υπέρ κατά απο... νομίζω ότι απορρίπτεται Παρακαλώ να ζητάτε έλεγχο αν θέλετε για να ξέρω τι να κάνω. Ελέγχουμε λοιπόν τη 438. Τέσσερα, 14 ε, της Επιτροπής ΕΜΒ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 54 447. Τροπολογία 447 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην σελίδα 56 και στην τροπολογία όχι, διορθώνει η πρόεδρος, σελίδα 55, συμβιβαστική 19. 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 458, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε διάφορες που έχουν καταπέσει. 463 στην σελίδα 57. 463. Ναι, ναι. Υπέρ κατά αποχές 464 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μάλλον πάμε στην 62. 480, τροπολογία 480. «482 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, ε, απορρίπτεται, 483 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 485 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα, αλλά μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Έχουμε χρόνο. We close the vote. And it is rejected. Απορρίπτεται. 488 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 Ήτρε υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 51 Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα περνάμε στην 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 498 7 4,97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4,98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4,99 υπέρ κατά ελέγχουμε την 4,99 ηλεκτρονικά. Στι της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24 κατά 20 υπέρ. 500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 28, 28, όχι, 29. Πού είναι 29? Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 507 υπέρ κατά Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 507. 508. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 ένβη υπέρ κατά αποχές γκρίνεται εγκρίνεται 31 31 υπέρ Πέντε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, περίμενετε. Διακόπτουν την Πρόεδρο. Τι θέλετε να ξαναψηφίσουμε την 514. Να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Τέλος. Απορρίπτεται. Εκτρά. Ντροπή κάποιον, ντροπή, ντροπή κάποιον. Βλέπω εγώ ποιοι ψηφίζουν και ποιοι, ψηφίζουν και ποιοι όχι. Και βλέπω και ποιοι, ποιοι ψηφίζουν κατά του ε, εισηγητή. 5-17 τώρα. 5-17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-19. Όχι, έχει καταπέσει. 521 υπέρ κατά, κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 24 κατά, 21 υπέρ. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 24 της Envy. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. is very difficult. And the votes. come on, still, yeah, yeah, now we can close. And if 24. 24 κατά προς 20 υπέρ απορρίπτεται. 5-22 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Έχουμε δύο τμήματα, ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5-2-4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εντάξει. 5-24 ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται. F33. 5-3-3. 5-3-3. Πάμε στην 533 λέει η πρόεδρος. 533 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εάν θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, να ελέγξουμε. Ναι. Άμα μου πείτε τσεκ, θα κάνω τσεκ.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 535. Του Μποτστινάρου. Can we vote? You, you found the... Τι έγινε, το βρήκατε να ψηφίσουμε. 5.35 υπέρ, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 5.39 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Ποιο είπε χωριστή και ψηφοφορία σε τμήματα. Όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Α, ακυρώνουμε την προηγούμενη ψηφοφορία και ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 539. Υπέρ. Κατά. Ποιες. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Δεύτερο τμήμα της 539 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 540 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση του 540. Επαλήθευση. Εγκρίνεται. Και τώρα Τώρα στη σελίδα 72, 553. Σε δύο τμήματα όμως. 553 στη σελίδα 72 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Πρέπει να το ξανακάνουμε γιατί είναι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Ένα μυστήριο πράγμα. 47 κάρτες είδαμε και ψηφίζουν μόνο 41. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως, ορίστε. Τώρα το τμήμα 2 του 553 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 554 υπέρ, κατά, αποχές, δεν απορρίπτεται, απορρίπτεται. 555 υπέρ, Κατά. Ποιες. Κάρα απορρίπτεται. 37 τραν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, επαλήθευση. Επαλήθευση για την 37. Ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 20-26. 5-56 υπέρ. Κατά. Ποιες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 559 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 στη σελίδα 76. Τραν 41. Βρείτε την μετά του κυρίου Σόνικ. Δεν τη βρίσκουμε φωνές. Α, έχετε άλλη σελίδα. Α, α λυπάμαι τότε. Τι να κάνουμε. Ποιος είναι υπέρ τέλος πάντων. Υπέρ τη 41 κατά 41 τραν με ταφ δηλαδή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 576 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ υπέρ, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 578 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 579 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 576 στην επόμενη σελίδα 586 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 592 υπέρ κατά χες. νομίζω ότι εγκρίνεται εγκρίνεται εγκρίνεται όχι, όχι, δεν ζήτησε κανείς απελευθέρωση, εγκρίνεται. 587 υπέρ. Α, Αποχές. Απορρίπτεται. Α, ήταν σε δύο τμήματα. 587 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όπως σαν να ήταν σε ένα τμήμα. Λοιπόν, 588 υπέρ για το πρώτο τμήμα, για το πρώτο τμήμα κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 μετά δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 589 πάλι σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 593 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 596 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 591 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε θα επαληθεύσω μεν ηλεκτρονικός αφού ζητάτε μπορώ να αρνηθώ δεν μπορώ Λείπουν πάλι μερικοί, λείπουν. Τέλο πάντων, απορρίπτεται. 43 υπέρ τη 43 κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 601 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 602 υπέρ όχι μα κατέπτε αν είχε εγκριθεί 601 απορρίφθηκε απορρίφθηκε 601 απορρίφθηκε όχι. Εγκρίναμε την 37 και λέει ότι 602 με 611 άρα καταπίπτουν. Ναι, αλλά εδώ στο 602 πρέπει να ψηφίσουμε. Το 602. «602 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». «603 υπέρ». Α, όχι, για πέστε μου, για πέστε μου. Α, 604 τώρα, 604 υπέρ 604 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 606 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 607 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 608 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 610 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 611 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 612 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 338-38 υπέρ κατά εγκρίνεται 614 υπέρ 614 614 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 615 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 616 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 621 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Όχι, επαλήθευση 621, γρήγορα, γρήγορα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Έληξε, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 627 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 629 υπέρ όχι ναι μα κοιτάξτε την 629 θα ψηφίσουμε τώρα και θέλω να σας τονίσω ότι η τροπολογία αυτή που είναι δική μου επιτρέπει στους άστεγους να ωφεληθούν από το Ταμείο Φεντέρ, το Περιφερειακό Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό. Η εισηγήτρια προτείνει καταψήφιση ενώ θα μπορούσε να είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, επαναλαμβάνω, για την καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων. Σα συστήνω να ψηφίσουμε υπέρ. Για αν θέλεις και εσύ να όχι λοιπόν να ψηφίσουμε. Ναι. 629. 629 υπέρ, κατά, χες, λυπούμε αλλά απορρίπτεται. 630 υπέρ, κατά, χες, απορρίπτεται. 631 υπέρ, κατά, οχές, εγκρίνεται. 632 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 635 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 634 υπέρ, 634, 33 ήταν πριν, 634 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση για το 634. Τι ωραία. απορρίπτεται πανηγυρικά 11 υπέρ 34 ε, κατά και τώρα τώρα 628 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 636 υπέρ 636 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 40 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα που είμαστε στο συμβιβασμό, όχι, 648, 648. επειδή είχε βρεθεί 40 καταλαβαίνετε. Α, Κωνσταντσα, καλά μας λες, 642 υπέρ. Λαμπέρ, 642 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα 648, 648 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 656 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εμπορύπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 659 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της 659 ξανά 22 υπέρ 24 ε, κατά απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Τώρα στη σελίδα 88 κάτω κάτω όπου λέει 60 ήτρε στην 89 ορισμένου. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επειδή εγκρίναμε τη 42 οι προσθήκες καταπίπτουν να μην με ρωτήσετε μετά γιατί δεν τις ψηφίζουμε. Λοιπόν. Τώρα που πάμε τώρα, συμβιβασμός 29. Συμβαστική 29, σε τρία τμήματα, σε τρία τμήματα, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν πάμε στη σελίδα 103 άρθρο 9 που λέει όπου λέει άρθρο 9. Εγώ δεν το έχω λέει πρόεδρος, δεν λέει άρθρο 9. Ποια τροπολογία είναι η 77. 77. Σε μερικούς είναι στη σελίδα 103. 103. Σε ποια σελίδα είναι αυτή η 50 τραν που λέτε κυριέ μου. 89, 50 τραν. 50 μετά, 89, 50 μετά, 50 μετά. 50 τραν λοιπόν, 50 τραν στην 89 κάτω κάτω. Κάτω κάτω, πρώτη τελευταία. Εκεί που λέει άρθρο 6 παράγραφος 3, 50 τραν. Υπέρ λοιπόν, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Και τώρα η 77. Στην 103 έχω εγώ το κείμενο λέει η πρόεδρος. Άρθρο 9, τίτλος. Τροπολογία 77. Λοιπόν, πάλι έλεγχος λόγω Γιάννου Ολμπριχτου ο οποίος μιλάει χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα. Σας κατευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, που άκουσε τι υπόθηκε. Τι ψηφίζουμε τώρα λοιπόν την 28 28 στη σελίδα 91 λέει όχι. Για ξαναπέστα τα Τι εννοεί τώρα, τι είναι. Πριν το συμβιβασμό 29 να ψηφίσουμε την 50 τράν 28 και 67 ήτρε. Αυτό ήθελα να πω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. 28 τράν υπέρ. Όχι, 28 ένβη, όχι τραν, 28 ένβη. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 67 ήτρε. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. Τώρα η 77, ε. Η 77. Η 77 ήτρε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 738 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 739 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 740 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 778 ή 378 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 745 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 746 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 747 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 748 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 750 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 751 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 752 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 753 υπέρ επαλήθευση για την 752 ηλεκτρονικός 752 απορρίπτεται 42 ψήφοι κατά, 3 ψήφοι υπέρ. 753 υπέρ, κατά, ποχές, απορρίπτεται. 754 υπέρ, κατά, ποχές, απορρίπτεται. 58 μετάφ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 755 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστικός 31, συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές, αποχές εγκρίνεται. 756 έχει καταπέσει, καταπέσει. 756 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 757 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 758 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 759 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 760 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 761 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 763 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 764 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 766 τώρα. Α και 65 αφού είναι η ίδια με την 64. 66 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, δεν κρίνεται, δεν Τώρα μετά 59, τραν 59, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 771 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 772 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 773 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 775 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 776 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 877 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 779 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 782 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 787 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 788 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54. Ε, 79 έχει καταπέσει. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56. Όχι, συγγνώμη. 790 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έχουμε τελειώσει. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε δύο ακόμα θέματα. Μετά την πρώτη ψηφοφορία θα πρέπει να συμφωνήσουμε για δύο πράγματα. Να δεχτούμε ότι αυτό που ψηφίσαμε μόλις είναι εντολή για τη διαπραγματευτική ομάδα στο να ξεκινήσει τη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Συμφωνείτε? ναι. Κάτε, κάντε κάτι. Φωνάξτε. Ηλεκτρονικά, ναι, ωραία. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, 37 υπέρ, 4 κατά. Και έπειτα το δεύτερο ερώτημα είναι αν η διαπραγματευτική ομάδα, ενώ όπως και στην προηγούμενη περίπτωση υπάρχει πρόεδρος, εισηγητής και ισχυώδης εισηγητές. Συμφωνείτε για αυτή τη διαπραγματευτική ομάδα? Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάνν Ολμπριχ θέλει να πει κάτι. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές που είναι έτοιμοι και που άλλαξαν την αρχική του θέση ε, αναζητώντα τη συμβιβαστική. Είμαι ευγνώμων. Τρει παρατηρήσει, αν μου επιτρέπετε. Πρώτη, πολύ συχνά πρότεινα να ψηφίσουμε μείον για κάτι που ήταν σωστό, αλλά που ήδη είχε προταθεί από το Συμβούλιο και ο Σκιώδης από κάθε πολιτική ομάδα έλαβε την πληροφορία για το ποια στοιχεία ρώτηνα να ψηφίσουμε όχι, ακόμα και αν ε, συμφωνώ, αλλά έχουν προταθεί από το Συμβούλιο. Ε, πολύ συχνά, δεύτερη παρατήση πολύ συχνά προτείνατε να αλλάξουμε τους θεματικούς στόχους και στο πρώτο γύρο σήμερα συμφωνήσαμε για τους θεματικούς στόχους ε, στο γενικό κείμενο. Προσπαθούσα λοιπόν να κάνω τη σύνδεση ανάμεσα στο γενικό κανονισμό και το δικό μου κανονισμό, ώστε να μην δημιουργηθούν αντιφάσεις ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο. Γι' αυτό και έγιναν όλες αυτές οι προτάσεις για αλλαγές ε, ε, θεματικών στόχων ε, μειωμένες. Έπειτα προσπάθησα να σημειώσω τα θέματα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν όπως η περίφημη τροπολογία της Καρή Μαντέλη για τους άστεγους. Δεν είναι τίποτα κατά των αστέγων, απλώς αυτό ήδη περιλαμβάνεται στο κείμενο που υπάρχει σήμερα για να, για να αποφύγουμε την κατάσταση ε, όπου μπορεί κάτι να μείνει εκτός. Δεν πρόκειται για σκάνδαλο, είναι απλά μια λογική ενέργεια για να αποφύγουμε τα υπερβολικά πολλά στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνουμε τώρα μια συζήτηση, δεν θέλω μάλλον να γίνει συζήτηση τώρα γιατί δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι κατάλαβα ο Μάρκος Πίπερ θέλει κάτι να πει. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ξαναπώ κάτι, να επισημάνω κάτι. Θα ήθελα και πάλι να επισημάνω ότι οι συμβασμοί έφτασαν στα χέρια μας εχθές το βράδυ. Και ο Γιάννη Όμπριχτ μας είπε επιλέξει δεν μπορείτε πλέον να αλλάξετε τίποτα στις συμβιβαστικέ προτάσεις. Δηλαδή, ο απλός βουλευτής στο μέλλον της Επιτροπής μας δεν είχε ούτε μία φορά την ευκαιρία να επέμβει σε αυτές τις συμβαστικέ προτάσεις. Αποτέλεσμα, αγαπητέ Γιάν πάνω από 25% των μελών δεν ακολουθούν αυτά που λέει ο κατάλογος ψηφοφορίας και αυτά που συνέστησες εσύ και παρακαλώ να το λάβεις υπόψη σου και να είσαι και δίκαιος και να συμπεριλάβεις και αυτούς που δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Και ε, επίσης πολλοί που υπερψήφισαν για να μην διακυβευτεί το όλο εγχείρημα δεν συμφωνούν. Έτσι όπως έγινε όμως ο χειρισμός ούτε διαφανής ήταν ούτε δίκαιος ε, πρέπει να πω. Κοιτάξτε, λέει η πρόεδρο, δεν θα γίνει συζήτηση. Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσω, λέει ο κύριο Όρμπριχτ, πώ θα γίνει προσπαθώ να είμαι πολύ διπλωματικός και να μην μπω στο μάρκος, ότι είναι καλό καμιά φορά να λέμε την αλήθεια. Έτσι καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Να είναι κανείς ειλικρινής. Οι συμβιβασμοί εστάλησαν σε όλα τα μέλη και τους σκιώδεις πριν από λίγες μέρες. Με τις ερωτήσεις. Συμφωνείτε να μπει η τροπολογία σας στο συμβιβασμό. Δεν ζήτησα κατά τμήματα ότι χωριστεί γιατί υπήρχε προθεσμία. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό μόνος συμβιβασμό που έκανα χτε το βράδυ, όπως το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ήταν κάτι που πρότειναν οι Γερμανοί συνάδελφοι και το συμφώνησαν με τους Γάλλους. Αν εσύ διαφωνείς, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά εμείς καταφέραμε να συγκεράσουμε πάρα πολύ διστάμενες απόψεις και οι δύο συνάδελφοι ήταν πάρα πολύ... Ε, συμβιβαστική σε πολύ επικοδομητικό πνεύμα. Αν αυτό επικρίνει, αφορά αυτό το συμβιβασμό. Είναι ο μόνο που άλλαξα χτε. Και δεν συμφωνώ. Και να μην λε στα μέλη τη Επιτροπή ότι αλλάξαμε κάτι νυχτιάτικα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ε, Τελείωσε η συζήτηση. Κυρία Ντελή, εντάξει, αλλά τελευταία. Ναι. Ένα λεπτάκι μόνο. Θέλω να σας καταστήσω όλους μάρτυρες. Είπε ο κύριος Όλμπριχτ ότι οι άστεγοι συμπεριλαμβάνονται και καλύπτονται από το συμβιβασμό και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αν αύριο στην επόμενη προγραμματική περίοδο δεν ενταχθούν οι άστεγοι, εκεί είναι που δεν έχουμε δικαίωμα να ψευδόμαστε. Ω και η συγκήτρια απέναντι στο Συμβούλιο θα φροντίσω αυτό το θέμα και σας το λέγω. Είναι κομβικό για μας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε οπωσδήποτε ότι η Επιτροπή μας δεν μπορεί να έθελο τυφλή απέναντι σε αυτή την αδιαφορία. Σας ευχαριστώ πάντως αγαπητοί συνάδελφοι για την υποστήριξη. Ευχαριστώ η Κωνσταντσε. Σα είπα δεν θέλω να γίνει συζήτηση. Ναι, εντάξει, παρακαλώ, πάρα πολύ σύντομα. Μετά από μια τέτοια συζήτηση δεν το θεωρώ σωστό να μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και οι άστεγοι άνθρωποι είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι και φυσικά ε, συμπεριλαμβάνονται και καλύπτονται από τα ταμεία. Τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά τώρα, υπερβολές, με πολιτικές θέσεις να τις κάνουμε αιχμή του δώρατος πάνω στην ψηφοφορία. With this we will move now to the next... Καλώς. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία που είναι του κυρίου Μποστινάρου, η έκθεση. Ελπίζω να είναι απλή. Δεν είμαι και σίγουρη. Αρχίζουμε. Συμβαστική 5. Ψήφι υπέρ τη συμβαστικής. Κατά του συμβιβασμού εγκρίνεται. Ο συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο συμβιβασμός 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ. Α, όχι, υπάρχει τροποφορική του εισηγητού, ο κύριος Βαστενάρου. Όντως, προτείνουμε να διαγραφεί από τις δραστηριότητες μέχρι τον αποκλεισμό και όλο το υπόλοιπο να παραμείνει ως έχει. Ωραία, όπως τροποποιήθηκε η 6 λοιπόν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 10 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ, Α, ε, γυρίστε σελίδα. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, εγκρίθηκε, συγγνώμη. Η 46. 8. Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές η συμβαστική εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 12 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 Envy υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 15 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 69 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 74 υπέρ. Αμέσως κάτω από το συμβιβασμό. 74. Κάτω από το συμβασμό 19 είναι. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία 77, το δεύτερο τμήμα ψηφί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 συμβιβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 συμβιβαστική δύο σελίδες πιο κάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 ή όχι. Απεριφθεί 16 της Τραν και 24 της Ένβη. Όχι. Α, ναι, αυτό εννοούσα, ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 91. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 92. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 93 ψηφοφορία κατά τμήματα ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 σε δύο τμήματα και ψηφίζουμε το δεύτερο υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 19 τράν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα αυτό τι σημαίνει, έτσι που το ψηφίσατε, καταπίπτουν τα παραρτήματα και πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις και διψηφίζουμε. ψηφίζουμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε πολλές σελίδες εδώ και δεν τα βρίσκω. Συμβαστική 1 στη σελίδα 23. Το έχετε εσείς. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 3. Ορίστε παρακαλώ. Να περιμένω. Το βρήκατε. Η τροπολογία 3 υπέρ Τρία του προπολογισμού υπέρ κατά Ψηλά τα χέρια, τα υπέρ. Ωραία. Εγκρίνεται. Για την τρία ρωτάω. Και εσείς σηκώσατε όλοι τα χέρια ψηλά. Υπέθεσα ότι εγκρίθηκε. Ο κύριο Βλάσσακ θέλει έλεγχο, το ελέγξουμε. Πέρας. Περίπου φτάνουμε στο πέρας, δεν κλείνουμε ακόμα, τώρα κλείνουμε. Πω, πω, κρίθηκε με μεγάλη διαφορά. Ε, οι δύο της ΙΤΡΕ είπε κατά άποχες. Τώρα δεν ξέρω τι κάνετε. Έλεγχος για τη δύο της ΙΤΡΕ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δεν έκλεισε ακόμα. Σχεδόν, περίπου, κλείνει. Απερίφθη. Η τροπολογία 4 του προπολογισμού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 5 ε, ψηφοφορία κατά τμήματα, τα δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 16 πρέπει να ψηφιστεί υπέρ κατά Έλεγχος για τη 16 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εμείς είμαστε υπέρ. Ε, υπέρ. 20 υπέρ, 23 κατά απορρίφτεται. Η τροπολογία εξ προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 2 προφορική, διαφωνεί κανείς με προφορική τροπολογία, όχι την ψηφίζουμε όπως τροπολογήθηκε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η τροπολογία 7 του προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Δύο μεταφορών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα... Πού Στην τέσσερα των μεταφορών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 5 των μεταφορών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ή μήπως έλεγχος για την πέντε. Αρχίζει τώρα ο έλεγχος. Για την πέντε των μεταφορών. Λάμπερτ, τι λέει το γουίπ εδώ. Α, υπέρ. is close and it's adopted 25 to 19. 25-19. Εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην 6 μεταφορών. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επτά μεταφορές. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 NV υπέρ κατά αποχές απορρίφθη. 8 τραν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 τραν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 σε 2 τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σχέδιο δεν το ψηφίζουμε, είπαμε, μόνο τις τροπολογίες. Βίκτορ, τελειώσαμε. Την ξεπετάξαμε την έκθεσή σου μέσα σε 10 λεπτά. Πριν πεις τίποτα, θέλω να πω τα εξή δύο εγώ. Ε, πρώτον, αυτό που ψηφίσαμε μόλις μπορούμε να το θεωρήσουμε ως εντολή για Βίκτορα και Σία για να μπορέσουν να πάνε να διαπραγματευθούν Συμφωνείτε, σηκώστε τα χέρια σας για να το πραγματικά ότι είστε υπέρ, ωραία. Ε, δεύτερον, για τη διαπραγματευτική ομάδα και πάλι είναι η πρόεδρος, ο εισηγητής και η σκιώδης. Συμφωνείτε με την ομάδα αυτή, τη διαπραγματευτική, όλοι υπέρ, πολύ ωραία, λαμπράκια σας ευχαριστώ και πολύ γρήγορα τώρα θα περάσουμε στο επόμενο.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 Να αρχίσουμε τώρα. Εντάξει, ακριβώς στις 5 θα τελειώσει. Ακριβώ. To say Dear colleagues, I am asked now by the colleague from the Regi eh, Secretariat. Οι συνάδελφοι από τη γραμματεία της ΠΕΡΙΦ ζήτησαν να μην λάβετε υπόψη το τελευταίο μήνυμα που σας έστειλαν, γιατί στις 2 και 4 μάθαμε ότι ο κατάλογος ψηφοφορία θα είναι ο ίδιος με τον χθεσινό με μία και μόνη αλλαγή και οι τροπολογίες 259 και 13 είναι ταυτόσιμες και οι 253 με την 257. You will see it in the vote. So if you understood, then it's fine. I did not, but I'm just not. I don't care. Αρχίζουμε λοιπόν. Με την μετάφοχτό, μετάφοχτό. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση της Ρίκας Μάνερ. Και υπάρχει κατάλογος ψηφοφορίας. Τραν 8 υπέρ. Μετά 8 υπέρ. Κατά. Όχι, επαλήθευση. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 101 101 υπέρ κατά απορρίπτεται 102 υπέρ κατά απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά απορρίπτεται 105 υπέρ κατά επαλήθευση για την 105 ε, 107, 107 απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά επαλήθευση για την 131 αλήθευση απορρίπτεται 27-17 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίθηκε, επαληθεύεται. 134 γρήγορα γρήγορα. Έλξε, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 3, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα Χριστέ μου πού να πάμε. 192 στη σελίδα 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω επαλήθευση για την 198 επαλήθευση απορρίπτεται τραν 17 στην επόμενη σελίδα α όχι όχι 207 πρώτα 207 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται 208 υπέρ κατά επαλήθευση για τη 208. Απορρίπτεται. Τραν, τραν 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 236 προφορική τροπολογία ε, ένα πρόβλημα, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 11, τραν 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 252 υπέρ, κατά, όχι, επαλήθευση για τη 252 αλήθευση απορρίπτεται 200 συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ κατά επαλήθευση για τη 263 απορρίπτεται 267 υπέρ 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 272 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 273 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 290 σε δύο τμήματα για το δεύτερο τμήμα υπέρ όχι το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά Ξανά ηλεκτρονικά 292. Απορρίπτεται. 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ κατά επαλήθευση 299. Εγκρίνεται. Κοντ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω επαλήθευση 312 απορρίπτεται 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 317 υπέρ κατά ξανά ηλεκτρονικά 317 17 απορρίπτεται 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 328 υπέρ κατά επαλήθευση την 328 ενεκρίθη 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 21 υπέρ κατά νομίζω εγκρίνεται νομίζω εγκρίνεται ελέγχουμε ξανά επαληθεύουμε την τραν 21 απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 331 υπέρ κατά θα την ξαναελέγξουμε And it's rejected. Απορρίπτεται. 333 υπέρ. 333 υπέρ κατά Πάλι δεν ξέρω, γιατί δεν ψηφίζεται και θα χρειαστεί να ξαναεπαληθεύσουμε την 333. Ψηφίζεται. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 346 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμού 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 349 Α, όχι, τη 40 πρώτα. 40. Υπέρ. Υπέρ. Αυτό το σκιασμένο. Υπέρ. Ξέρει τι λέει ο Φρανκ. 40 είπαμε. Μα επιμένει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, 40 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 348. Α, καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. 349, 349 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Ξανά. 349. Τι δύσκολα πράγματα. Προλαβαίνουμε. Α, προλαβαίνουμε. Ένας σοσιαλιστής δεν ψήφισε. Ο Κύριλο, ή ήρθε παραπάνω ο Κύριλοφ. Αν θέλετε να μπορέσει να ψηφίσει και ο Ευγένη, πρέπει κάποιος άλλος να μην ψηφίσει. Τώρα εντάξει, τώρα εντάξει, τώρα εντάξει. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 350 υπέρ, κατά, ποχές, απορρίπτεται. 351 υπέρ, Λαμπέρ, κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Μα δεν φαντάζεστε τι δύσκολη επιτροπή που είστε για ψηφοφορία, ρε παιδιά. 351 επαλήθευση. Άντε ρε παιδιά, μόνο 37 ψηφίζουνε. Απορρίπτεται. 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμού 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 354 354 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κοντ 7. Ελέγχ 7. Ο, ναι, ελέγχ 7 υπέρ. Κατά, όχι, απορρίπτεται. 356 είναι κανεί κατά επειδή είναι προφορική, όχι υπέρ. Κατά, 356, 256. κατά αποχές εγκρίνεται. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές. 358 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 359 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απερίφθη αλλά θα επαληθεύσουμε την 359. Τι θα κάνουμε Λαμπέρ. απορρίπτεται. 360 υπέρ, 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 361 υπέρ κατά επαλήθευση. Απορρίπτηκε Κοντ 8, Ελέγχο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε νομίζω. Εγώ βλέπω το αφεντικό άμα είναι αυτός υπέρ. 362 υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Ε, επαλήθευση, μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται για δύο ψήφους. Ελέγχ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχ όχι 364 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε δεν διαμαρτύρεται καν μια 42 Περ. κατά αποχές εγκρίνεται 43 Πώς 366 στην δεν θα το δεχόμουν αυτό, σήμερα είμαι καλή, λοιπόν θα ελέγξουμε την 366, ορίστε. Δεν ψηφίζουν όλοι, παιδιά. 21 υπέρ, 19, ε, κατά 19 υπέρ, ορίστε. 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 368 υπέρ 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 23 υπέρ τι μπλοκ μπλοκ και τις τρεις της τραν μαζί εντάξει και οι τρεις της τραν μαζί λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Α, έχουν και άλλες τράνε εδώ. Λοιπόν, 26 με 28 όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 269 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 29 υπέρ. Α, μαζί, μαζί, μαζί, ναι. 29 μέχρι και 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Το σκεπτικό, α, το σκεπτικό τώρα, το σκεπτικό δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Προϋπολογισμό 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, προϋπολογισμό 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το σκεπτικό 1 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται. Κοντ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Όχι, 51, 51. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπό λέξη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική για το σκεπτικό 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπόλεπτα λεπτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική για το 10 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται Τραν 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Επαλήθευση, επαλήθευση, επαλήθευση. Εσείς θα μετανιώσετε για την 73. Α, απορρίφθηκε με δύο ψήφους παραπάνω. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά επαλήθευση για το 78 επαλήθευση απορρίπτεται Προϋπόλ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 σε τμήματα, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ ο, επαλήθευση του 82, επαλήθευση για την 82. Απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τραν 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τραν 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ υπέρ ξανά κατά έλεγχος γιατί είναι 86 Πέρες απορρίπτεται 24-17 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Μάλλον τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται αν δεν κάνω λάθο. Προπολογισμό 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 90 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Και τώρα 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ υπέρ κατά Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Στην 93 είμαστε. Έτσι δεν είναι. Όχι, 94. Την 94 ελέγχουμε. Ανοίγω την ψηφοφορία. Την 94 ελέγχουμε αυτή τη στιγμή. Πέρας. 27 κατά, 13 υπέρ, άρα απερίφθη 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά ε, κοντ 2 της ε, λέγω του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί ε, Επαλήθευση. Εντάξει, εντάξει, 99. we do with uh, the uh, so what we do tomorrow 2020 2020 20 ισοψηφία, άρα χάσαμε. Ε, θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να το λέει ο Μιγγέλ, κάτι θα ξέρει. Πέρασε. Τώρα τι να πω. Α, για τη διαπραγματευτική εντολή. Ναι, ναι, τα ίδια ε, με προηγουμένω. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό που ψηφίσαμε θα θεωρηθεί διαπραγματευτική εντολή για την ομάδα. Όλοι συμφωνούν, μάλιστα. Δεύτερον, από ποιον θα απαρτίζεται τώρα. Πρόεδρος, ε, εισηγήτρια και σκιώδεις εισηγητές. Και αυτό θα πρέπει να το εγκρίνει ως απόφαση η Επιτροπή. Μου λέει ο Μιγγέλ ότι η τελευταία ψηφοφορία είναι τόσο μικρή και τριανταφυλένια που μπορούμε να τη διεκπαιρεώσουμε τώρα αμέσω. Αλλά να αποφασίσει ο Γιώχιμ Τσέλερ αν θέλει να ψηφίσουμε το θέμα του ή So you don't know how to vote? Τι, δεν ξέρετε πώς θα ψηφίσετε. Εμείς πάντα ακολουθούμε την πρόεδρο, λέει ο κύριος Βανίστερόι. No, no, so, so what is What is... very short,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 Are you ready to? Can we start the vote? Yeah, okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Τσέλερ. Η τροπολογία 42. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Εάν 11 υπέρ. Είναι για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Ε, κανείς δεν διαφωνεί με την προφορική. Η τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Ναι. 47 υπέρ. Κατά. Απόχες. Και αυτή νομίζω. Αν θέλετε έλεγχο, ελέγξουμε. Τι έλεγχο θέλετε. Για τη 47, ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Να κοιμάστε ήσυχοι, μην έχετε ανησυχία το βράδυ δηλαδή. Χάνουμε κόσμο, δεν ψηφίζετε. Τώρα. 22 υπέρ 16 κατά ε, εγκρίθηκε. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έχουμε το 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 όπως τροποποιήθηκε προφορικά και δεν διαφωνεί κανείς τη ψηφίζουμε έτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 στο 2 τελική σκέψη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 έτσι δεν είναι, καλά τα λέω. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ 2. 2. Του. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά η επαλήθευση για την 5. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. 24 υπέρ 17 κατά. Ποια τελευταία είπαμε η 5. Και τώρα 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά... Νομίζω ότι εγκρίνεται, εντάξει. 40 υπέρ τι θέλετε, έχω για ποια. Για την 9. Καλώ. Αρχίζει το ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 26 υπέρ 15 κατά. Πάμε στην 40 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελειώσαμε! μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτό που μόλις ψηφίσαμε μπορεί να αποτελέσει διαπραγματευτική εντολή για τον Γιάχεμ Τσέλερ και τους υπολείπου. Ωραία, συμφωνείτε. τη δεύτερη ερώτηση, τα γνωστά, η πρόεδρος και τα λοιπά, η διαπραγματευτική ομάδα. Πρόεδρος, ε, εισηγητή και σκιώδη. Και αυτό το εγκρίνουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο επόμενο θέμα, η έκθεση του Όντρεχ Βλάσακ. Ορίστε. Nobody. Dear colleagues, I would like to... Συνάδελφοι, παρακαλώ να ανακοινώσω κάτι. Ακούστε το κι αυτό. Επειδή δεν χρειάζεται αύριο να ξεψηφίσουμε γιατί είχε προβλεφθεί μένα αλλά δεν χρειάζεται αύριο αντί για ψηφοφορία στις 10.30 θα συνεχίσουμε την ημερήσια μας διάταξη. Καλύτερα αντί να γίνει τώρα διάλειμμα, να γίνει τότε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα τελειώσουμε νωρίτερα αύριο. Παρακαλώ λοιπόν να το λάβετε υπόψη σας. Δεν θα έχει ψηφοφορίες αύριο, αλλά θα συνεχίσει η κανονική εργασία της Επιτροπής μας. Και τώρα συνεχίζουμε το 14, το 14 του κυρίου Βλάσακ, γνωμοδότηση για τον ορίζοντα 2020 έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εισαγωγικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις ψηφοφορίες. Είμαι πολύ ευτυχής που καταφέραμε να τελειώσουμε και γρηγορότερα από ό,τι νομίζαμε. Ήταν τεράστια η πρόκληση και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και συνεισηγητές. Διότι ήταν πολύ βοηθητική. Και τώρα περνάω στην ε, έκθεση. Μιλάμε για το ορίζον 2020. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα και όλες οι τροπολογίες είχαν στόχο να οθήσουν την ανάπτυξη και την συμμετοχή των περιφερειών, πόλεων και τοπικών κοινοτήτων που δεν αντικατοπτρίζεται αρκετά στην ε, πρόταση ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κρατημέλη να αυξήσουν αυτές τις δραστηριότητες στα λειτουργικά τους προγράμματα για την έρευνα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Εγώ πιστεύω πως το Horizon 2020 θα πρέπει επίσης να λάβει σοβαρά υπόψη την γεωγραφική διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηρίξει τις ερευνητικές πρωτοβουλίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Πράγμα που κατά τη γνώμη μου θα ενισχύσει την περιφερειακή διάσταση της ε, ερευνητικής πολιτικής και των επιστημών. Γι' αυτό θα ήθελα να δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση στην ε, διακρατική διάσταση του προγράμματος. Πιστεύω λοιπόν πως η έκθεση αυτή, αυτή η γνωμοδότηση και όλες οι τροπολογίες θα πρέπει να σας ε, δώσουν ε, κίνητρο για να ασχοληθείτε με αυτή την έκθεση. Γι' αυτό θα ήθελα να πάρετε εσεί το λόγο. Εγώ πολύ προσεκτικά θα σημειώσω όλα σα τα σχόλια και αν έχετε το χρόνο. Καλό θα ήταν να μου τα στείλετε και ηλεκτρονικά για να τα συμπεριλάβω στην τελική εκδοχή του κειμένου μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στου σκιώδει. Σαλβατόρε Καρόν είναι ο πρώτο σκιώδη. Και εγώ Καρόνα. Α, συγγνώμη, ο Μυροσλάβ είναι εδώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρέπει να πάρει το λόγο πρώτος ο Μυροσλάβ. Ή όχι, όχι. Ας σας αφήσουμε εσά κύριε Καρόνα. Απλώς ξέχασα ότι είναι εδώ ο Μυροσλάβ Νικολάσης που είναι επίση και Έλεγα και εγώ ότι συμμερίζομαι το γεγονός ότι η πρόταση της Κομισιόν για το ορίζον 2020 είναι μια καλή βάση, ένα καλό σημείο κίνηση για να ορίσουμε τις δραστηριότητες της, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, <clears throat> το θετικό στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι η δομή σε τρεις πυλώνες, η ολοκλήρωση σε ένα μόνο πρόγραμμα ολόκληρη αλυσίδας καινοτομίας από την έρευνα μέχρι την αγορά, η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης σε μια απόπειρα απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Αυτά είναι τα σημαντικά και ισχυρά σημεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Όσον αφορά εμάς ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, θα πρέπει να διορθώσουμε νομίζω Αυτή την ε, προσέγγιση του κανονισμού όσον αφορά την μεγαλύτερη συμμετοχή, την ε, πιο ξεκάθαρη ενίσχυση δηλαδή της πτυχής των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι πολύ σημαντικές έτσι ώστε να προχωρήσει στεναρά όλο αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω λοιπόν πως ένα από τα βασιμελιώδη σημεία είναι, θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ορισμός ενός ρόλου για τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές και αυτό σε ε, συνδυασμό με μεγαλύτερο συντονισμό του προγράμματος Horizon 2020 και όλο την υπόθεση των διορθωτικών ε, ταμείων. Καλύτερη σύνδεση λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημαντικά ταμεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Λείπει ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να υπογραμμίσουμε. Μια σαφής δηλαδή μνήμα στις ε, επενδύσεις στις ερευνητικές ε, στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και της ε, συντήρησης και της διατήρησης του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού ε, κληροδοτήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει πιο έντονα και πιο αποφασιστικά να το αντιμετωπίσει και το πρόγραμμα Horizon 2020. Θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες σχετικά στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάσικ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σχολιάσω αυτό το ενδιαφέρον έγγραφο που συζητούμε. Πράγματι, ζητώ, επιζητώ συνεργασία και με τον εισηγητή και με τους άλλους συναδέλφους. Με τον συνάδελφο Βλάσακ μέχρι τώρα η συνεργασία μας ήταν πολύ θετική και γι' αυτό θα είναι για μένα πολύ ευχάριστο και στο μέλλον να συνεργαστώ μαζί του για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα, ιδίως αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητος. Πρέπει να σκεφτούμε ποια θέλουμε να είναι η μελλοντική κατεύθυνση των... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι ζητούμε περισσότερη ανάπτυξη για τη βιώσιμη ζωή της οικονομίας μας αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Το πρόγραμμα Horizon 2020 μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και θα μπορούσε να βελτιώσει και τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παγκοσμίω. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα στήριξης που βασίζονται στον κύκλο της ε, καινοτομίας και της έρευνας. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το Horizon 2020 θα χρειαστεί να επιμείνουμε ιδιαίτερα στις διαδικασίες που εγκυώνται τη χρηματοδότηση ορισμένων βασικών προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της ζωής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής και για μένα αυτό είναι η εκκίνηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πρόσβασή τους σε ενωσιακά ταμεία. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχει και, ένα άλλο, και μια άλλη σημαντική πτυχή για την ευρωπαϊκή έρευνα που είναι ότι γίνεται αυτή τη στιγμή διενεργείται σε διάφορους τομείς στη βιολογία, στην ιατρική και η ποιότητα της ευρωπαϊκής έρευνας πρέπει να συμβαδίζει με τα, τις δεοντολογικές και ηθικές αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι βασικές ηθικές αρχές στηρίζονται στις συνθήκες και στη χάρτα των θεμελιωδών καθώς και σε όλα τα άλλα βασικά νομικά μας κείμενα. Όταν μιλάω για ποιότητα εννοώ ότι Πρόκειται και για υψηλή ποιότητα ηθικά πρότυπα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ιδιότερα συνάδελφοι τα ηθικά αυτά πρότυπα που εμφαίνονται στα νομικά κείμενα και που τα αναφέρει πολλές φορές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα λαμβάνονται πάντοτε υπόψη από όλα τα κράτη-μέλη. Η χρηματοδότηση λοιπόν της έρευνας, της έρευνας λέω που φέρνει σε επαφή όλα αυτά τα προβλήματα με τις ηθικές αρχές πρέπει να συμβαδίζει με αυτές. Όταν δεν συμβαδίζει είναι απαράδεκτη. Και θα ευχαριστώ. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Χάιντερούδερ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα τον εισηγητή, διότι στις προτάσεις του έλαβε υπόψη ακριβώς αυτό για το οποίο είναι αρμόδια η Επιτροπή μας. Και βέβαια το πρόγραμμα Horizon 2020 περιλαμβάνει πολλά στοιχεία γιατί είναι ο διάδοχος του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Αλλά το θέμα είναι οι δικέ μας προτεραιότητες εδώ στην Επιτροπή μας. Εκεί θα πρέπει να επιτροθούμε και να μην πλατιάσουμε. Γι' αυτό θεωρώ την πρότασή του πάρα πολύ καλή για τον περιφερειακό χαρακτήρα που τονίζει και τον διαμεθοριακό και το υποστηρίζω. Η μόνη πρόταση που θα είχαμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη η συμπερίληψη κοινωνίας των πολιτών, η ε, αρχή της εταιρική σχέσης και αυτό να μπει παρακαλώ και θα κάνουμε μικρές βελτιωτικές ε, τροπολογίες. Κατά τα άλλα υποστηρίζουμε απολύτως τη γραμμή του εισηγητού και τον ευχαριστούμε. Και νομίζουμε ότι είναι καλή συνεργασία μας εκεί. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι πρόεδρος. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Κουπρέκης, θέλετε να πείτε τίποτα. Sorry. Ξέχασα τον κύριο Βανίστεροι. Okay, uh, I Πάλι νόμιζα ότι είχα καθυστερήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται στο τσάκ ήρθα. Λοιπόν, όντως αυτό είναι ε, πώς να το πω, από τα σημαντικότερα προγράμματα. Όταν μιλούμε για συνέργειες, τι θα πει αυτό, μεταξύ των διαφόρων μέσων περιφερειακής πολιτικής, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα με τη θεματική τώρα ε, πλέον επικέντρωση που έχουμε. Και βρισκόμαστε σε μια θέση όπου θα μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα Horizon 2020 στο μέλλον. Πριν από λίγο ψηφίσαμε μόλις. Αυτό το θέμα της εδαφικής συνεργασίας. Και φέραμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για να υπάρχει ακριβώς αυτή η συνεργασία των περιφερειών στο δρόμο προς την αριστεία. Στο παρελθόν Ορισμένα προγράμματα ε, που είναι στο σημερινό 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, τον κάτοχο ας πούμε του Horizon, του Horizon έχουν βγει. Αλλά υπάρχει ένα ερευνητικό δυναμικό ε, ε, σε αυτά τα προγράμματα που έχει τώρα πλέον ενσωματωθεί στην εδαφική συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα αυτό, διότι το πρόγραμμα Horizon έχει ένα βασικό κριτήριο. Την αριστεία. Ε, ο καλύτερος καθηγητής. Από, να μην πω τώρα πανεπιστήμιο, δεν έχει σημασία από πού θα έρθουν οι καλύτεροι καθηγητές. Ε, διασυνδέονται και συνεργάζονται και επιλέγονται. Αλλά υπάρχουν τόσες πολλές περιφέρειες που έχουν το δικό τους δυναμικό και μπορούν να καλύψουν διάφορους τομείς τεχνολογίας για ε, την κλιματική αλλαγή, για την ενεργειακή μετάβαση, ε, για θέματα με μεγαλύτερο κοινωνικό προσανατολισμό, αλλά αυτή ακόμα δεν είναι ε, στο ζενή, θα πούμε, της αριστείας. Και αν θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη, δεν αρκεί να έχουμε ένα θαυμάσιο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα ή τον ορίζοντα, 2020, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση αυτή την καινοτομία να τη μεταφέρουμε στην πράξη. Τα ερευνητικά αποτελέσματα να μεταφραστούν σε εφαρμογές, ε, σε νέα υλικά, σε νέες μεθόδους, ε, να γίνουν πραγματικότητα. Αν συγκρίνουμε, ας πούμε, την Ευρώπη με τις Ηνωμένε Πολιτείε, Έχουμε εξαιρετικά Ινστιτούτα και γνώση, αλλά υπολοιπόμεθα ε, στην ταχύτητα μεταφοράς αυτής της καινοτομίας και στην αλυσίδα για την υλοποίησή της. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία που σήμερα στην εδαφική συνοχή δεχτήκαμε και εγκρίναμε τη δυνατότητα κάποιων περιφερειών που δεν είναι ακόμα στο top της αριστείας, σε πάση περιπτώσει, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Και αυτό ονομάζουμε κλίμακα αριστείας. Και το έχουμε και στο γενικό ε, κανονισμό και στο ΕΤΠΑ. Είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον 1% και μέχρι και 10% να μπει σε αυτό το στοιχείο της συνεργασίας στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γιατί τα λέω αυτά όλα. Διότι είναι πραγματικά το αποτέλεσμα της συνεργασίας που έχουμε ε, με το έργο μας εδώ και το πρόγραμμα ορίζον. Ίσως, Όλτριχ ε, Βλάξακ, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και αυτά τα στοιχεία στη δική σου πρόταση για να πούμε ότι δεν είναι απλώς το πρόγραμμα Horizon 2020 που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να περάσουμε σε μια νέα φάση για στενότερη συνεργασία και να δημιουργήσουμε όντως ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας για πιο μακροπρόθεσμα, να έχουμε ιδιαίτερες περιφέρειες που να εξειδικεύονται, όπως και σήμερα συμβαίνει εξάντεκ των προτέρων ε, να υπάρχει αυτή η αιρεσιμότητα με την ευφυή e e λεγόμενη εξειδίκευση. Ε, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το βήμα αυτό και κάπου να τονίσουμε περισσότερα και να δείξουμε περισσότερα από αυτά που μόλις ψηφίσαμε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Γιατί όταν δεν τα λες αυτά τα πράγματα, σε αγνοούν. Συγγνώμη που σας τρώω το χρόνο, αλλά τι να κάνω. Ήθελα να τα πω. Έπρεπε να βάλω και εγώ το λιθαράκι. Ευχαριστώ. Is a special session, you know, after. Σήμερα είναι ειδική σύνοδος. Είναι εδώ κάποιος από την Επιτροπή, κύριος Κορπάκης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, so, Δημήτρη Κορπάκης, European Commission, Digital Research and από την Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Κοινοτομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα χρήσιμά του σχόλια. Πιθανότατα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλε τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί, διότι υπάρχουν ε, κάποιε που δεν. Θα ήταν εύκολο να εφαρμοστούν όπως αυτή για την ε, εδαφικοποίηση αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εφαρμογή του προγράμματος Horizon 2020 και σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο κ. Βανίστερ Ρόι θα ήθελα να θυμίσω ότι οι υπηρεσίε της Κομισιόν από την έρευνα και την καινοτομία και την περιφερική πολιτική έχουν συνεργαστεί πολύ στενά ε, στο επίπεδο των κανονισμών και έχουμε φτάσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με την ευφυή e διοικευσή ε, και τον σχετικό όρο, αλλά και με τις ρήτες όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση, όπου οι περιφέρειες πρέπει να δαπανίσουν συγκεκριμένα ποσά για θέματα ανταγωνιστικότητας και έρευνας και γενοτομίας. Να σας θυμίσω ότι έχουμε φτιάξει ένα κοινό δελτίο που έχει κυκλοφορήσει στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου υπό το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, το Δελτίο 28 που δίνει πολλές λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τη ε, σύνδεση ανάμεσα στο ορίζοντα 2020 και τα διευθυντικά ταμεία και πώς αυτά θα γίνουν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορπάκη. Ε, κύριε Βλάσακ, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνέβαλαν στη συζήτηση. Φυσικά σημείωσα τα σχόλιά σας. Συμφωνώ απόλυτα με πολλά πράγματα που υπόθηκαν εδώ. Δεν σημαίνει μόνο μείωση του διοικητικού φόρτου, και βελτίωση της πρόσβασης σε ενισχύσεις και δημοσιονομικά μέσα, αλλά πρόκειται και γι' αυτό που είπε ο κύριος Βανίστελ Ρόι, δηλαδή τη διάδοση νέων γνώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας να τεθούν σε εφαρμογή. Η σύνδεση δηλαδή της έρευνας με την πράξη, ιδιαίτερα στις περιφέρειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, συμφωνώ με τα όσα ε, ε, ε, είπαν και οι σκιώδεις εισηγητέ ε, πρέπει, και το είπε και η κυρία Ρίλε, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να διανύμουμε τη στήριξη αυτή παντού. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, συγκεντρώσουμε τη χρηματοδότηση και να χρησιμοποιήσουμε τις ε, συγκεκριμένες δυνατότητες στην Ευρώπη και στις περιφέρειες. Και εδώ υπάρχει πεδίο για συνεργασία ανάμεσα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Θα προσπαθήσω να δω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει, ποιες είναι οι τροπολογίες αυτές για να αποφύγουμε τα προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε τελική συμβιβαστική που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχόλια σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 16 Ιουλίου το μεσημέρι. 16η Ιουλίου, ναι. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι το υπαρθμό 15, ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ο κύριος Βλάσακα έχει και πάλι το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη από τον Λαμπέρτ που μιλάω τόσο πολύ. Γιατί ο Λαμπέρτ είναι ο εισηγητής φυσικά μαζί με την Κωνσταντσα και προσπαθώ και εγώ να παίξω τον ίδιο σημαντικό ρόλο με εκείνον. Η οικοδόμηση των διευρωπαϊκών δικτύων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ακόμη όμως έχει ορισμένα εκκρεμή προβλήματα χρηματοδότησης, επαρκούς ύψους χρηματοδότησης. Δεν θέλω όμως να το ζητήσουμε τώρα, δεν θέλω. Θέλω απλώς να τονίσω ότι προσπάθησα στην έκθεση γνωμοδότησή μου να πω μόνο τα εξής. Μεγαλύτερη ελαστικότητα για τις χώρες μέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σπουδαίο γιατί χρειάζεται, μου φαίνεται, η συζήτηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών των χωρών μελών να γίνει. Τα προκαθορισμένα προγράμματα δεν πρέπει να θεωρούνται σαν κάτι τελειωτικό και το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να είμαστε να είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες συγκεκριμένων χωρών μελών. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν γίνεται οι τοπικές αρχές να είναι υπεύθυνε για προγράμματα που ξεπερνούν τις δικαιοδοσίες τους διότι δεν διαπραγματεύονται εκείνες τα προγράμματα και άρα αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τέλος, τέλος λέγω, μπορεί ήδη να τα έχετε δει αυτά στα, στις επιστολές που σας έστειλα. Πιστεύω ότι πρέπει όταν εξετάζουμε τα μεμονωμένα προγράμματα, όταν εξετάζετε εσείς τα, που εκείνα που ενδιαφέρουν τα κράτη σας, να μου λέτε και μένα τι συμβαίνει. Και εγώ για την Τσεχία έκανα ορισμένες συγκεκριμένες ε, παραπομπές σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αν θέλετε να βάλω και δικές σας να μου τις στείλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε και πάλι. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις συζήτητες. Ο πρώτος, ο κύριος Ματούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, βεβαίως, πρέπει να αρχίσουμε με την ιδέα ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι ένα ολοκληρωμένο ε, πανευρωπαϊκό δίκτυο που θα πρέπει να ενσωματώνονται όλα τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό που εξακολουθεί να υπάρχει, ιδιαίτερα στις πρόσφατα εισηγμένες χώρες. Επίσης, ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια απλοποίησης. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα πρόσδεκτο. έχουμε φτιάξει και αυτόν τον οδικό χάρτη πρόσφατα για τον ευρωπαϊκό χώρο με έμφαση σε ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών όσον αφορά τους πόρους και πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που φτάνει μέχρι το 2030 ή και το 2050. Κάποια σημεία αντιμετωπίζονται γέννη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καταρχήν το σημερινό διευρωπαϊκό δίκτυο χωλαίνει στις, διευρω... στις, στις ε, περιοχές συνοριακές όσον αφορά την ποιότητα αλλά και την ύπαρξη υποδομών για τη σύνδεση ανάμεσα στα κρατημέλη. Επίσης, ε, η, υποδομές μεταφορών θα πρέπει ε, να είναι και ε, διατροπικές. Πρέπει να βρούμε δηλαδή διατροπικές συνδέσεις. Ε, κόμβους, να κατασκευαστούν κόμβοι, λιμένες, αερολιμένες, οι οποίοι λείπουν, ιδίως στα πιο νέα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών μέχρι 60% και να ανταποκριθούμε και στην ανάγκη για διαλειτουργικότητα σε πολλούς τομείς. Είναι λοιπόν σημαντικό στην ανάλυση μας να τα εξετάσουμε όλα αυτά ο εισηγητής μίλησε για χρηματοδότηση, θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Δεν είναι απλά θέμα συνοχής με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι Έχουμε τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη επίσης στην πολιτική μου ομάδα, το ΕΛΚΑ, Έχουμε συζητήσει αυτή την ανάγκη για, μελλοντικό, για το μελλοντικό διευρωπαϊκό δίκτυο στο τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, γιατί εδώ παίζουν ρόλο κλειδί οι διάδρομοι μεταφορών. Υπάρχει προστιθέμενη αξία που θα πρέπει να προκύπτει από τα έργα σε αυτό το τομέα. Και θα πρέπει να είναι επίση σαφέ ότι πρόκειται για προγράμματα μεταφορών που χρειάζεται τη στήριξη των κρατών μελών. Αν σκεφτούμε τι επιπλέον προσπάθειε που θα πρέπει να καταβάλουν τα κρατημέλη. Νέα πρόκληση για τα κρατημέλη που εν γέννη τείνουν να προτάσουν ε, τις εθνικά ή τοπικά περιφερειακά προγράμματα ή έργα, ενώ τώρα η πρόκληση είναι να στηριχθούν τα κρατημέλη και να κινητοποιηθούν, να παροτρινθούν ώστε να φτάσουν σε προγράμματα διασυνοριακά, ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε ένα δίκτυο μεταφορών το οποίο να μπορεί γρήγορα να προωθηθεί ώστε να, προωθηθεί, ώστε να προωθηθεί ταυτόχρονα και μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα παλιά και στα νέα κρατημέλη από Ανατολή σε Δύση καθώς και να συνδεθούν τα νησιά με την υπηρετική Ευρώπη. Θέλουμε την εσωτερική αγορά, αλλά εσωτερική αγορά και για μεταφορές. Και θα επαναλάβω τα συγχαρητήριά μου προς τον εισηγητή. Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για αυτό το θέμα, όταν θα δούμε και την τροπολογίες που θα έχουν κατατεθεί και βεβαίως να εξισορροπήσουμε τα <clears throat> δικαιώματα των τοπικών αρχών και περιφερειών στον τομέα. Θα έχουν περισσότερες ευθύνε από ό,τι στο παρελθόν και να δούμε και τον κατάλογο των διαδρόμων που είναι ενδεικτικό θα πρέπει να, να συζητήσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως η περιοχή των Άλπαιων καθώς και οι απομονωμένες νησιωτικές περιοχές όπου θα πρέπει να δούμε την ε, διαλειτουργικότητα ε, και να συντονίσουμε την ανάπτυξη για τις διασυνοριακές υποδομές. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς, λέει κύριος Κύριλο Φωτή, συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή κύριο Βλάσακ ότι η ε, πρόταση του κανονισμού αποτελεί καλή βάση για τις μελλοντικές ε, διαδικασίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης ε, των υποδομών που έχουν διευρωπαϊκή σημασία. ορίζουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει νέα θετικά στοιχεία που βασίζονται σε εφιστάμενες οδηγίες κατευθυντήριες γραμμές, ας πούμε. Ε, μια δίκτυη προσέγγιση για το δίκτυο υποδομών, ε, μεταφορών που να ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις γραμμές και ένα βασικό δίκτυο ε, οδικό στους αυτοκινητοδρόμους. Επίσης, αξίζει το κόπο να μιλήσουμε για τους διαδρόμους, για καλύτερη κατασκευή αυτού του βασικού κεντρικού δικτύου καλύτερη συνεργασία, καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων των κρατών μελών που ε, θα υποδεχθούν αυτούς τους διαθρόμους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν συνδέσεις και είναι ε, μεγάλες ε, οι στενοποί και τα προβλήματα ιδιαίτερα σε κόμβους τα προβλήματα αυτά πρέπει να λυθούν και θα βοηθήσει αυτό, θα ενισχύσει σίγουρα ε, την εδαφική συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των περιφερειών και θα τονώσουν και την οικονομική ζωή και την κοινωνική συνοχή. Και αυτό νομίζω είναι από τις βασικές αρμοδιότητές μας. Έτσι θα βελτιωθούν ε, οι συνδέσεις με γειτονικέ χώρες, θα σπάσουν τα σημεία συμφόρησης και ε, οι μεγάλες ροές και οι ε, επιβατικές και ε, οι εμπορευματικές θα προωθηθούν. Όπως είπε και η σα, αυτή είναι πραγματική προστιθέμενη αξία. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα ολοκληρωμένο σύστημα και δίκτυο χωρίς διακοπές και με καλύτερη πρόσβαση. Ορισμένες από τις τροπολογίες στο σχέδιο νομοδότησης ε, συμπληρώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη σκοπιά της δικής μας Επιτροπής. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που δεν λέγω ότι δεν τις έχουμε σκεφτεί αρκετά, αλλά νομίζω ότι υπερβαίνουν λίγο τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Και είμαι βέβαιος ότι οι τροπολογίες 10 με 17 του κυρίου Βλάσεκ είναι πολύ χρήσιμες, αλλά έχω την αίσθηση ότι ε, μήπως δεν είναι ακριβώς η αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής, γιατί αν μπούμε σε αυτά τα χωράφια, γιατί μας ζητάει να προτείνουμε αντίστοιχε τροπολογίες, νομίζω ότι υπερβαίνουμε ε, τις δικές μας αρμοδιότητες και δεν είναι πάρα πολύ επικοδομητικό αυτό. Αν θέλετε το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή του συντάκτη της νομοδότησης και θα κάνω κάποιες τροπολογίες για θέματα διασυνοριακά και περιφερειακά, καθώς επίσης και την ευθύνη των Ευρωπαίων Συντονιστών. Γενικά κάνουμε πολύ καλή δουλειά και ο εισηγητής κάνει καλές ε, προτάσεις και καλές ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίας. Ε, Αν δούμε την πρόταση της Επιτροπής και τους στόχους της, και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Επιτροπή μας. Ε, κατά τα φαινόμενα μπορούμε να εκφράσουμε θετική γνώμη, γιατί φαίνεται να είναι μια ισορροπημένη θέση, δηλαδή θέλει να φτιάξει σύγχρονες μεταφορές, συνδεδεμένες, διαλειτουργικές, κανείς δεν έχει τίποτα εναντίον. Όταν γίνεται λόγος για έργα προτεραιότητας επί τη βάση του κοινού συμφέροντος και αξιοποίηση αυτών που έχουν προσθέμενη αξία, επίσης δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, θετικά αξιολογούμε την πρόταση. Όμως ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι αν στόχος της Κομισιόν Περιφερειακής, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι να λάβει υπόψη αυτές τις διαφορές ε, και τις διαφορετικές ε, προοπτικές ολοκλήρωσης με τα διάφορα, τις διάφορες περιφέρειες φοβούμαι ότι θα πρέπει να αποκαλύψω και σε πολλούς συναδέλφους ότι θα απογοητευτούμε τα μάλα καταρχήν διότι δεν θα καταφέρουμε να αγγίξουμε τίποτα ούτε σε σχέση με τη χαρτογραφία ούτε σε σχέση με τους διαδρόμους ούτε σε σχέση με οποιαδήποτε δυνατότητα αλλαγής. Και αυτό το λέω γιατί προέρχομαι από, την Επιτροπή Μεταφορών. Εκεί ήδη Ήρθαμε σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε, να εντάξουμε, αλλά εκεί περισσότερο οι κυβερνητικές πιέσεις, οι πιέσεις του Συμβουλίου είναι αυτές που κυριαρχούν. Εκεί καθορίζονται οι, γραμμές, οι χάρτες, τα σημεία κτλ. Τούτου λεχθέντος και μαζί με τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε για να μπορέσουμε να υποβάλουμε τροπολογίες, ε, θεωρώ πως έχουμε καθήκον να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα ώστε να επιβεβαιώσουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας σκοπιά, ότι δηλαδή θέλουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ε, δαφών, των περιφερειών, ώστε να τονίσουμε αυτήν την ανάγκη επαφή με τις περιφέρειες και βέβαια όχι φτιάχνοντας ένα ευχολόγιο με και δρομάκια που μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι έχουν ε, κοινό συμφέρον και γενικό, είναι μάλλον και για κοινό όφελος, αλλά να μιλήσουμε για τις αρχές όπως την ανάγκη ένταξης εντό του κεντρικού δικτύου συνδέσει με περιφερειακέ ζώνε ή με νησιωτικέ ζώνε, Πρόεδρε. Νομίζω πω αυτό είναι καθήκον μα. Τώρα, στη συνέχεια, Εξαρτώμαστε από την Επιτροπή Μεταφορών και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε την ίδια αντιμετώπιση, ότι δηλαδή θα απορρίπτουν τις προτάσεις που έρχονταν από τις διάφορες επιτροπές τη στιγμή που ασκήσαμε τη δική μας ε, αρμοδιότητα να αξιολογήσουμε τις προτάσεις που έγιναν επί των ε, κανονισμών που εγκρίναμε σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση, αλλά ως πράσινοι έχουμε αρκετές αντιρρήσεις σχετικά με τις τροπολογίες που προτείνει η γνωμοδότηση του κυρίου Βλάσακ. Είμαστε υπέρ της συμμετοχής των περιφερειών και της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών για λόγους διαφάνειας, ολοκληρωμένης προσέγγισης σε θέματα μεταφορών και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης ο κανονισμός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών είναι καλή ευκαιρία για να μετασχηματιστεί το μοντέλο των μεταφορών προς, μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση συνδέοντας επιμέρους πολιτικές για να πετύχουμε την οικολογική και οικονομική βιωσιμότητα. Α μην ξεχνάμε, οι μεταφορέ συνδέονται και με άλλε πολιτικέ. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να ανταποκριθούμε καλύτερα στι δεσμεύσει και του στόχου Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την προστασία τη βιοπικιλότητα, για την ανάπτυξη μεταφορικών κλάδων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, αλλά συμβάλλουν στην βιώσιμη ευημερία των τοπικών κοινωνιών και την πράσινη οικονομία. Ένα τέτοιο επαναπροσδιορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στι μεταφορέ σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των υφιστάμενων επενδύσεων και έργων μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των περιορισμένων έτσι και αλλιώς οικονομικών πόρων μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης. Είμαστε αντίθετοι να στρέφεται η χρηματοδότηση κυρίως σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και γιατί έτσι η Ευρώπη συνεχίζει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο και ταυτοχρόνως συνεχίζεται η επιβάρυνση ατμόσφαιρας και της υγείας των πολιτών συνολικά η χρηματοδότηση για αυτοκινητοδρόμους στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουμε δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30%. Να δοθεί λοιπόν προτεραιότητα στη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών για πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα, όπως το τρένο, η δάτινη δρόμη, οι συνδυασμένες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων και των ποδηλάτων. Αυτό σημαίνει ότι το 70% των χρηματοδοτήσεων πρέπει να στηρίξει παρόμοιες μορφές επιδιώκουμε την αποθάρρυνση χρήση γιοταχή αυτοκινήτων και φορτηγών για λόγους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και για λόγους υγείας. Αλλά για να πετύχουμε μια τέτοια πολιτική χρειάζεται να βελτιωθούν υποδομές συνολικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το τρένο, ποδήλατο, ακόμα και το περπάτημα. Μην ξεχνάμε και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μονοπατιών. Η βελτίωση υπαρχουσών διασυνοριακών συνδρομικών συνδέσεων και η επέκτασή του, εκεί που δεν υπάρχουν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ιδιαίτερα στα Βαλκάνια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει συνολικότερα σχέσει καλή γειτονία, αλλά και στην ενίσχυση οικονομικών συνεργασιών μεταξύ των χωρών. Έμφαση πρέπει να δοθεί στι συνδυασμένε μεταφορέ, δηλαδή μεταφορέ που συνδυάζουν διαφορετικά μέσα, που ελαχιστοποιούν τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου και το θόρυβο, καθώ και του κινδύνου ατυχημάτων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη διαχείριση Υποστηρίζουμε μια ουσιαστική επαναξιολόγηση προκειμένων έργων στη βάση του κόστους και της ωφέλειας για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σήμερα που αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα από την κρίση και υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση των κοινωνιών. Για παράδειγμα, στη χώρα μου την Ελλάδα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της χρήσης, πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι πραγματικά χρήσιμη οικονομικά και κοινωνικά ε, και οικολογικά βιώσιμη όλοι οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που δεσμεύουν άμεσα ή έμεσα ένα μεγάλο ποσό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων την ίδια στιγμή που απαξιώνεται ο σιδηρόδρομο. Θα ήταν πιο σωστό να, ανακατε... να ανακατευθύνουμε μέρο τουλάχιστον των πόρων σε πιο βιώσιμα μεταφορικά έργα, όπω για παράδειγμα το μετρό στην Αττική και Θεσσαλονίκη, το τραμ, δίκτυα ποδηλατόδρομων, που θα αναζωογονούσαν την οικονομία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και θα δημιουργούσαν πολύ περισσότερε θέσει εργασία, αλλά σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει μια πίεση να ολοκληρωθούν τα έργα, κυρίως από μεγάλε κατασκευαστικές εταιρείε από τη Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία. Η στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι επίση σημαντικό να έχει μια συνολική προσέγγιση και να μην αντιμετωπίζει κάθε έργο χωριστά. Ε, πιστεύουμε ότι το άρθρο 42 για την περιβαλλοντική προστασία πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ε, χρειαζόμαστε την περιβαλλοντική διάσταση την ενσωμάτωση αναλύσεων κόστους ωφέλειας και την ενίσχυση συνοχής μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών αλλά και επιμέρους προγραμμάτων αν θέλουμε μεταφορές να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής ένωσης για το 2020 αλλά και για να καλύψουν με αποτελεσματικό και οικολογικά αποδεκτό τρόπο τις ανάγκες των πολιτών. Προτείνουμε λοιπόν ο στόχος σημείας του εξωτερικού κόστους, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, να αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργων. Μια και προέρχομαι και από νησιωτική περιφέρεια, θέλω να τονίσω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών πρέπει να επεκτείνονται και στα νησιά, αλλά και σε ρακοτυγμένε περιοχέ. Οι υδάτινοι δρόμοι και οι θαλάσσιε συνδέσει, ακόμα και για μικρέ αποστάσει, είναι όχι μόνο αποτελεσματικέ, αλλά στην περίπτωση των νησιών σχεδόν ο μοναδικό τρόπο σύνδεσή του με τι υπόλοιπε περιοχέ και με την Ευρώπη. Α μην ξεχνάμε ότι τη χρήση αυτών των συνδέσεων δεν την κάνουν μόνο οι νησιώτες αλλά την κάνουν Ευρωπαίοι πολίτες από όλες τις χώρες του κόσμου, από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Θεωρούμε επίσης ότι οι διαδρομές του γύρω Βέλο για το ποδήλατο πρέπει να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Οι προτάσει Κομισιόν για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αλλά και του θορύβου πρέπει να διατηρηθούν και δεν συμφωνούμε με την πρόταση να αλλάξουν. Η μείωση στην πηγή του θορύβου από τα τρένα αλλά και το ERTMS θα πρέπει να μείνουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Τέλος, χρειαζόμαστε πιο σαφή ορισμό των όρων συνδέσεις που λείπουν, διασυνοριακός και στενοπή, bottlenecks. Ε, και ήθελα να ευχαριστήσω, θα καταθέσουμε βέβαια τις αναλυτικές μας προτάσεις μέσα από τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, is there Commission who wants to... Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κανείς το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή για την έκθεσή του και για τα σχόλια από τους σκιώδεις που όλοι τόνισαν νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν καταφέρνει τον τετραγωνισμό του κύκλου δηλαδή επικεντρώνεται στις υποδομές και την εσωτερική αγορά ενώ παράλληλα διασφαλίζει την συνοχή στην Ευρώπη. Δύο σχόλια έχω να κάνω για την έκθεση. Πρώτον, ε, και τα δύο μάλλον συνδέονται με τον κύριο στόχο της πρότασής μας που ξεπερνάει την απλή συμπερίληψη των νέων στόχων στα διευρωπαϊκά δίκτυα γιατί συμπεριλαμβάνει και την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τώρα η ενωσιακή επικράτεια είναι πολύ μεγαλύτερη. Η πολιτική των TEN-T, των διευρωπαϊκών δικτύων, είχε σημειώσει αρκετές επιτυχίες, αλλά μία από τις αδυναμίες της ήταν ότι δεν υπήρχε επαρκής και καλή διακυβέρνηση και σαφέστερος καθορισμός των προτεραιοτήτων που ενδιαφέρουν πολύ τους πολίτες. Πώς καταφέραμε λοιπόν αυτόν τον τετραγωνισμό που σας έλεγα. Βασικά προμηθεύσαμε ένα πλαίσιο που προβλέπει οι χώρες μέλη και τα όργανα της Ένωσης να δεσμευθούν μέχρι το 2030 να έχουν δημιουργήσει αυτό το βασικό δίκτυο που να καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική αγορά και να διασφαλίζει και maximum προστασία του περιβάλλοντος με παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών. Εξ ολόκληρη επαναλαμβάνω την επικράτεια της Ένωσης. Αυτή η βασική προσέγγιση υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο και κατά τις προκατασκευαστικές φάσεις της εξέτασης της πρότασής μας και γενικά εγκρίθηκε και από τους Υπουργούς Μεταφορών τον περασμένο Μάρτιο. Επομένως, η δέσμευτη αυτή για το 2030 συνδυάζεται με την ευελιξία που απαιτείται και που χορηγείται στις χώρες μέλη για την εφαρμογή των προτύπων, για τις εξαιρέσεις, όλες τις ευελιξίες που απαιτούνται για να μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει αυτό το βασικό δίκτυο. Δεύτερο στοιχείο είναι η αυξημένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στην πρότασή μας βλέπετε ότι βασιζόμαστε στην ευρωπαϊκή μεθοδολογία που έγινε σε συνεργασία και με τους υπουργούς και η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στις χώρες μέλη και στην Κομισιόν κατά την προετοιμασία της πρότασης να κάνουν, επέτρεψε να κάνουν δύσκολες επιλογές. Αλλά βέβαια η διαδικασία αυτή επειδή στόχευσε τις κύριες προτεραιότητες διασφάλισε τη δυνατότητα των χωρών μελών πράγματι να πραγματοποιήσουν το βασικό δίκαιο μέχρι το 2030. Αν λοιπόν κατατεθούν τροπολογίες θα πρέπει να δοκιμαστούν αυτές με βάση την μεθοδολογία αυτή για να μην υποθούν πράγματα που τελικά δεν ανταποκρίνονται στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Τρίτον δε στοιχείων, η διάδρομη του βασικού αυτού δικτύου που θα υπάρχουν από την αρχή γιατί η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται φυσικά σε αυτούς, θα χρειαστεί χρηματοδότηση για ολόκληρο το σύστημα των TEN-T, αλλά θα δοθεί σημασία στους διαδρόμους για να υπάρξει μεγαλύτερος και καλύτερος συντονισμός. Uh, Παρ' όλα αυτά Σταματάω μάλλον εδώ και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής και τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ κύριε Βλάσακ. Θέλετε να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ε, δεν θέλω να επαναλάβω τους βασικούς στόχους των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και βέβαια θα πρέπει να ε, λύσουμε τα σημεία συμφόρησης. Αυτό ισχύει για λιμένες, αερολιμένες ή και για κάποιους κόμβους και σταυροδρόμια ε, όπως και τα διασυνοριακά δίκτυα. Αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά η Επιτροπή μας συνεισφέρει από τη σκοπιά της περιφερειακής πολιτικής και των περιφερειακών φορέων. Αυτό είναι το δικό μας πρίσμα. Και έχουμε το δικαίωμα να επηρεάσουμε ε, το κείμενο με τη δική μας ε, τοποθέτηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνεργαστούμε με ε, τις ε, πολεοδομίες φεριπίν. Αυτό είναι αρμοδιότητα ε, τοπική και όχι κεντρική ε, για τα μεγάλα έργα και για τις μεγάλες χαράξεις και γραμμές. Υπάρχουν και μελέτες αντικτύπου περιβαλλοντικού που είναι αρμοδιότητα εθνικών υπουργείων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται συνεργασία όλων αυτών των εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Και ε, πρέπει να σας πω ότι ίσως χρειάζεται να εξηγήσω τις ε, τροπολογίες μου σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι όλοι μας, εδώ τους βουλευτές, έχουμε μια ιδιαίτερη πατρίδα. Ο καθένας ξέρει στην ιδιαίτερη περιφέρεια του τι γίνεται και έχει την ευθύνη να εκπροσωπεί ε, όσο μπορεί την περιφέρειά του και τα συμφέροντά της και αυτά να ε, τα προτείνει στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα στοιχείο αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Βεβαίως και γνωρίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε λεπτομερείς λύσεις για τα διάφορα προβλήματα. Από την άλλη όμως ε, δεν μπορούμε και να τα αποφεύγουμε. Αν θέλουμε να τα λύσουμε πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική επιχειρηματολογία για να μπορέσουμε να πείσουμε και την καθήλη ε, αρμόδια επιτροπή που προκειμένου είναι η Επιτροπή Μεταφορών. Ένα τελευταίο. Αυτά τα θέματα του περιβάλλοντος όπως είναι ο θόρυβος κλπ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι Ό,τι φράγμα και να βάλεις, ε, τείχος για να σταματήσεις ε, την ηχορύπανση από αυτοκινητοδρόμους ή διάφορες γέφυρες ή, τούνελ και σύραγγες για να περνούν οι βάτραχοι Φερρυπίν, είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ε, γιατί είναι θέματα που επιβαρύνουν ιδιαίτερα το κόστος κατασκευής ενός αυτοκίνητου δρόμου. Και όταν μιλούμε για διευρωπαϊκά δίκτυα, χρειάζεται ένας προγραμματισμός, ένας σχεδιασμός. Δεν μπορεί σε μια χώρα ένα χιλιόμετρο αυτοκίνητο δρόμου να κοστίζει ένα χι και να επιβαρύνεται υπερβολικά το κόστος επειδή είναι ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Και δεν θα πρέπει να υπάρξουν μεγάλες αποκλήσεις γενικά λόγω αυτού. Ένα τελευταίο. Θα πρέπει ε, τα έργα αυτά, τα διευρωπαϊκά, να είναι αηφόρα, βιώσιμα, ε, αλλά σε ό,τι αφορά τις πόλεις και τις αστικές συγκοινωνίες δεν ξέρω ε, κατά πόσο επαρκούν τα κονδύλια για να αφιερωθούν και εκεί. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι η διασύνδεση της Ευρώπης και όχι πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης της πόλης. Αυτά τα ε, ε, ολίγα θα λάβω υπόψη τη τροπολογίες και χαίρομαι για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την προθεσμία υποβολής τροπολογιών η οποία είναι στις 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Τελευταίο θέμα τη σημερινή συνεδρία ο Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτος 2013 όλα τα τμήματα. Είναι δική μου έκθεση, γνωμοδότηση μάλλον, και θα ήθελα να την παρουσιάσω στη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και στη συζήτηση για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την εντολή για τον τριμερή διάλογο, έτσι και στη σημερινή συζήτηση για το σχέδιο γνωμοδότηση τη ΡΕΤΖΙ σχετικά με τον Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2013, το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Η πολιτική συνοχή είναι το κύριο και πιο κατάλληλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόληση, αντιμετωπίζοντα με ακρίβεια τι επενδυτικέ ανάγκε των περιφερειών και συμβάλλοντα την πραγματική μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την επίτευξη κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση καλωσορίζω την αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 1β κατά 3,3% και την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 11,7% σε σύγκριση με τον προπολογισμό του 2012. Η τελευταία αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιοριστεί η αύξηση των προσεκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση της Επιτροπής αφορά αυστηρά το 2013 και λαμβάνει ως δεδομένο ότι οι ανάγκες πληρωμών από παρελθόντα έτη θα έχουν καλυφθεί και ως εκ τούτου οποιαδήποτε απόκληση από αυτή θα οδηγήσει σε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών. Η Επιτροπή στη διαμόρφωση των προβλέψεών τη για τον προπολογισμό έχει αποτιμήσει τι ανάγκε, λαμβάνοντα υπόψη τι διατάξει τα ανώτατα όρια των πιστώσεων από τι δημοσιονομικέ προοπτικέ 2007-2013 και τη διοργανική συμφωνία και έχει ευθυγραμμίσει όλα τα αριθμητικά δεδομένα με τι σχετικέ αποφάσει και διατάξει Επομένω, το μοναδικό θεσμικό όργανο που διαθέτει τι σχετικέ πληροφορίε για να έχει τη γενική εικόνα των δημοσιονομικών αναγκών όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Σύμφωνα με τη θέση τη Επιτροπή Προπολογισμών του Συμβουλίου, που υιοθετήθηκε στι 5 Ιουλίου και αναμένεται να εγκριθεί σε επίπεδο COREPER, σήμερα και στο τέλο του μήνα από το Συμβούλιο των Υπουργών, το θεσμικό αυτό όργανο έχει προβεί για μία άλλη φορά σε οριζόντιε περικοπέ. Κατά συνέπεια, Ακολουθώντας την τακτική των προηγούμενων εισηγητών, προτείνω οι περικοπές του Συμβουλίου να ακυρωθούν και να επαναφερθούν τα ποσά που αρχικά προτάθηκαν από την Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού. Τέλο, επί του διαδικαστικού, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να σα υπενθυμίσω ότι μαζί με την Πρόεδρο έχουμε αναλάβει την εντολή να υποβάλουμε τα πιλωτικά έργα, τι προπαρασκευαστικέ δράσει ή και τα μέτρα τεχνική βοήθεια που έχουν συμφωνηθεί από τι πολιτικέ ομάδε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, Κανείς και ο εισηγητής θέλει το λόγο. Κρέλ. Παρακαλώ, η κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας υποστηρίζω στην γνωμοδότησή σας, Ρίτα. Ε, σήμερα το πρωί είχαμε την Κυπριακή Προεδρία και συζητούσαμε και ακούσαμε τον κύριο Γκοντμάνης που μίλησε για αυτά τα θέματα των υποχρεώσεων πληρωμών και θα πρέπει ακριβώς στην Περιφερειακή Επιτροπή ε, πολύ σιγά ακούμε ζητήματα απορροφητικότητας και μας mm. προσάπτουν ότι τα κράτη-μέλη δεν απορροφούν τα κονδύλια. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά όταν έχεις κάποια προγράμματα που τρέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί το Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να δώσει αρκετά κονδύλια για τις πληρωμές, ε, τότε δεν επιτρέπονται αυτά τα λένε και δυνατά και μεγαλόφωνα γιατί είναι πολύ κακή η κατάσταση. Και αν το Συμβούλιο δεν ε, πιστεύει τα ίδια του τα αριθμητικά στοιχεία και τα αμφισβητεί, πού θα πάμε. Γι' αυτό υποστηρίζω ρητά και οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις πληρωμών να επανέλθουν στο 11, πόσο ήταν ε, στη γνωμοδότησή μας και ελπίζω το Συμβούλιο πραγματικά να το καταλάβει, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς και να ε, χρηματοδοτήσει αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Βανίστεροι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με την Κωνστάτσα. Στο παρελθόν τα ακούμε αυτά συνέχεια. Λες και δεν το είχαμε ποτέ συζητήσει. Μα το έχουμε συζητήσει και στο γενικό ε, κανονισμό. Συμφωνώ απολύτω με την Κωνσταντσε Κρέλ. Κοιτάξτε τι κάνουμε τώρα. Ζητούμε να υπάρχει αρκετό χώρος για τις ε, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών που πρέπει να είναι στο 11,7%. Αλλά στην πρακτική τι γίνεται. Τσεκούρι από το Συμβούλιο και από την πείρα που έχουμε των περασμένων ετών θα πρέπει να πω ότι είναι τρελό αυτό το πράγμα. Από τη μια κάνουμε τους υπολογισμούς με τα διάφορα κονδύλια που επιστρέφουν αναπορόφητα, όχι τόσο από εμά, αλλά ε, πηγαίνουν ε, Στου κρατικού κορβανάδε και δεν λένε και ποτέ ευχαριστώ κατά τα άλλα, έτσι, εμπαρόδο. Και 2%, 2 του ευρωπαϊκού προπολογισμού επιστρέφει στα κρατικά ταμεία. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λογαριασμοί και των περιφερειακών προγραμμάτων και δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε αυτά. Είναι σχιζοφρένεια αυτό που συμβαίνει. Και θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο πολύ περισσότερο και να τους πούμε δεν μάθατε ακόμα. Άμα παίρνετε κάθε χρόνο 2% και 2,5% πίσω και τα εγγράφετε στον εγγρατικό σας προϋπολογισμό και μετά για τα επόμενα έτη δεν είστε διατεθειμένοι να δώσετε τα λεφτά. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα πληρωμών μετά και στο τέλος της προγραμματικής περίοδου που θα είναι το 13 του χρόνου ε, οξύνεται ακόμα, επιτείνεται το πρόβλημα σημειώνω ότι έχουμε και απλήρωτους λογαριασμούς ακόμα από το 11, έτσι, κληρονομήσει στο 12. Και τώρα από το 12 θα τους μεταφέρουμε στο 13. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα. Ε, χώρες που έχουν και ε, δηλώσεις αξιοπιστίας έρχονται το Δεκέμβριο μετά διαπραγματεύσεις και όλα αυτά που κάνουμε με το Συμβούλιο και πέφτει μεγάλη περικοπή και το Δεκέμβριο έρχονται οι δηλώσεις τους. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Λεβαντόφσκι το έχει πει επανειλημμένα και σε εμά άλλωστε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εμένα, θα μπορούσαμε να είμαστε και οξύτεροι και να πούμε ότι αν έχουμε αυτό το περιθώριο, εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι. Όχι, να πούμε να έχουμε αυτό το περιθώριο. Αλλά αν η κατάσταση συνεχιστεί, ε, θα έχουμε μεγάλο έλλειμμα. Και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες λέμε αναλαμβάνουμε υποχρεώσει. Πρέπει να τι πληρώσουμε. Αυτό το καταλαβαίνει ο πολίτη. Άμα πα να του πει όμω ότι έχω τον προπολογισμό του 2013. Αλλά μειώνεται, ξέρει, ο προπολογισμό. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουν οι πολίτε. Ξέρω εγώ, παγώνει και όλα αυτά τα πράγματα, περικοπέ, ε, γιατί και στα κράτη-μέλη είναι δύσκολη η κατάσταση και οι πολίτε οι ίδιοι δυσκολεύονται και καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται περικοπέ. Αλλά το μουτζούρι το κληρονομούμε εμεί ω κοινοβούλιο. Και σε εμά ρίχνουν το φταίξιμο και μα λένε ότι ορίστε, εσεί θέλετε να αυξήσετε το προπολογισμό. Μα αυτό είναι η ίδια η συστηματική. Αν δεν είναι κάποιο πρόθυμο να εξηγήσει το προπολογισμό ότι έχουμε βρει παιδιά λογαριασμού και πρέπει να του πληρώσουμε. Και ε, τα περασμένα χρόνια είχαμε ε, πλεονάσματα και τα δώσαμε πίσω στα κράτη-μέλη. Έτσι διωγγώνεται το πρόβλημα και φταίει το Συμβούλιο. Δεν ξέρω. Ίσως αυτά θα πρέπει να μας τα εξηγήσει κάποιος από την Οικονομική Επιτροπή. Αλλά να λέμε όλη την ιστορία και όχι πάντα ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά και όλο να στέλνουμε λεφτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε και να το υπερασπιστούμε. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσα να επιμείνω κι άλλο ε, σε αυτό το θέμα, αλλά άμα ε, μας ξεφύγουν και οι πολίτες και δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε. Χάνουμε και την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω, ίσως να το διατυπώσουμε καλύτερα. Εγώ θα ε, ε σας υποστηρίξω στο αίτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάγκα, παρακαλώ Σας ευχαριστώ. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διάφορα τμήματα και μόνο ένα από αυτά αποκαλείται, τυλοφορείται Επιτροπή. Είναι το τμήμα 3. Υπάρχει το τμήμα του Κοινοβουλίου, το άλλο του Συμβουλίου, το ΔΕΚ τα κτλ. Φυσικά, σήμερα εξετάζουμε το τρίτο τμήμα της Κομισιόν που περιλαμβάνει και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία που αφορούν εμάς, στο τμήμα δηλαδή που, είναι, αφορά το κοινοβουλικό. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποια σημεία εδώ. Υπάρχουν μεταφρασμένα κείμενα τα οποία παίρνουμε ε, μαζί μας στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι μεταφρασμένα όλα τα τμήματα στις γλώσσες μας. Οι μεταφραστές κάποιες φορές μεταφράζουν τα κάποια τμήματα του κειμένου σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Δεν γίνεται λοιπόν ε, δουλειά έτσι όμως. Γιατί μπορεί να τύχει πολύ σημαντικά κομμάτια που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στη γλώσσα μας να μην είναι έτοιμα στην ώρα τους. Και αυτό δεν μας βοηθάει. Έπειτα έχει συμβεί επανειλημμένως διάφορα θεσμικά όργανα να μεταφράζουν τα έγγραφά τους από τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες και έχει τύχει να χρησιμοποιούν και εξωτερικούς ε, συνεργάτες μεταφραστές. Αυτά όμως τα θεσμικά όργανα δεν έκαναν καν την προσπάθεια να δουν αν υπάρχουν μεταφραστές σε άλλο θεσμικό όργανο που θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά αυτή, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν εκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα. Δεν ξέρω ποια επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το θέμα των μεταφράσεων, αλλά ίσως και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Well, thank you very much. I thank all... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τα ενδιαφέροντα σας σχόλια και προσβλέπω στη δική σας και σας ευχαριστώ μόνο για την υποστήριξή σας. Πριν κλείσουμε τη σημερινή συνεδρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι και επίσης η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για το σχέδιο προπολογισμού είναι η 27 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ όλους.